Good afternoon. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ε, επόμενη συνεδρίαση, δεν τελειώσαμε ακόμα. Την τρίτη το απόγευμα θα γίνει η μεγάλη μας ακρόαση για την ψηφιακή ατζέντα. Μεγάλη υπόθεση για την Επιτροπή μας αλλά προς το παρόν περνάμε στην πέμπτη μας ενότητα. Αλλά τους επόμενους μήνες ε, θα έχουμε ακόμα πιο πολλή δουλειά. Εν περιπτώσει, εξαιρετικά σημαντικό θέμα τώρα. Δημόσια κρόαση με θέμα λύσης διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιε διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και του πολίτε. Γνωρίζετε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Θέλω να καλωσορίσω τους ομιλητές μας και να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος της Επιτροπής Ήτρα που δεχτήκατε να συμμετάσχετε σε αυτή την ακρόαση. Μας τιμά αυτό. Χρειαζόμαστε πάντα συμβουλές από τους επαγγελματίες. Ορισμένοι από εμάς είμαστε επαγγελματίες, ο καθένας στον κλάδο του. Και μοιραζόμαστε και ευθύνες και για την ψηφιακή ατζέντα στις χώρες μας χρειάστηκε να το χειριστούμε αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε εσείς τι έχετε να μας πείτε. Και οι επιτροπές ΙΝΚΟ και ΛΥΒΕ γνωμοδοτούν για θέματα της ακρόσης αυτής και τα μέλη τους έχουν προσκληθεί βεβαίως να παρευρεθούν. Δεν ξέρω μπορεί να, είστε παρόντες, να είναι παρόντες στη συνέχεια ορισμένα μέλη. Οι οι συντάκτες νομοδότησης, ΙΜΚΟ και ΛΥΜΠΕ ε, έχουν προσκληθεί. Ο, συγητής, ο συντάκτης νομοδότησης της ΙΜΚΟ θα έρθει, της ΛΥΜΠΕ δεν μπορεί. Μια μισή ώρα έχουμε προβλέψει, στις 4.30 κανονικά πρέπει να έχει τελειώσει αυτή η ακρόαση. Θα ήθελα καταρχάς να παρακαλέσω από πλευράς μας να μας κάνει μια παρουσίαση ο συγητής και μετά τη ΣΥΜΚΟ, ο συντάκτης νομοδότησης, μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα ενημερωθούμε για ε, δύο ε, μελέτες ε, περιπτώσεων που έχουν γίνει, μία στην Πολωνία, η άλλη στην Πορτογαλία. Ο Κάρλος Ζωρίνιο είναι ο εισηγητής μας. Να σας διαβάσω και πάλι τον τίτλο «Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις και τους πολίτες». Εξυγχρονισμό του δημοσίου τομέα ουσιαστικά είναι το σύνθημά μα. Έχετε μέσα στο λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω τι ευχαριστίε μου για την ευκαιρία που έχουμε να κάνουμε αυτή την ακρόαση. Και είναι ένα ζήτημα σημαντικό, όπω και η ακρόαση αυτή άλλωστε. Θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων εδώ. Οπότε, στα σχόλιά μου δεν θα παρουσιάσω την έκθεση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο θα κάνω είναι να επισημάνω κάποια από τα σημαντικά ζητήματα. Όπω είπε ο πρόεδρο, η ψηφιακή ατζέντα είναι ένα από τα βασικά ζητήματα και κινητήρια δύναμη μαζί με την ενεργειακή μεταβολή που θα δημιουργήσουν κάποια ελπίδα στην Ευρώπη για ένα πιο ανταγωνιστικό και δίκαιο μέλλον με ανάπτυξη και δουλειές. Αυτό ακριβώ έχει κάποια προτεραιότητα η επένδυση σε αυτόν τον τομέα, άρα είναι σημαντική για τους στόχους της ευελιξίας και βεβαίω για να χρησιμοποιήσουμε και άλλο μέσα. Η διαλειτουργικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ πέρα. Γιατί Εάν τα θεμέλια σε ένα σπίτι είναι σάπια, μετά ό,τι βλακάκια και να βάλουμε το σπίτι θα πέσει. Αυτό είναι λοιπόν το βασικό σημείο αναφοράς. Εάν το φτιάξουμε σωστά, το πρόγραμμα θα είναι σωστό. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν πρέπει να πετύχει δύο πράγματα. Συνέχεια με τα προηγούμενα προγράμματα αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προβλέψει και τεχνολογικές αλλαγές, ζούμε σε καιρούς με αλλαγές, οπότε δεν μπορούμε να χάσουμε την ευκαιρία αυτή να ευθυγραμμίσουμε το πρόγραμμα με τις συνθήκες που έχουμε. ψηφιακή ατζέντα έμοιαζε κάπως ε, τεχνική, αλλά τώρα μοιάζει κάπως πιο πολιτική. Κάποιες από τις παλαιότερες ε, πρωτα... κάποιες από προτάσεις μου, που ελπίζω να στηρίξουν οι συνάδελφοι, ε, ήταν, έγιναν δεκτές από τους σκιώδεις συζητητές Και βεβαίως θα δείτε το πώς ακριβώς ε, θα διαμορφωθεί η πολιτική ατζέντα. Γιατί πρέπει να δούμε εδώ πέρα τι γίνει με το ψηφιακό αυτό θεματολόγιο για τα επόμενα δέκα χρόνια. Οπότε πρέπει να μεταλλευτούμε τα όσα είχαμε πει στο παρελθόν με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, να υπάρξει κάποια μεγαλύτερη ενημέρωση και τις ε, δυνατότητες ε, που δίνει. Δεν ε, είναι δυνατόν απλά να λέμε λόγια. Πρέπει να εμπλακούμε πιο πολύ με τους πολίτες, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία να ευνοήσουμε τις ε, συνεργασίες και να προσπαθήσουμε να μην αποτύχουμε σε αυτό το θέμα κλειδί που είναι η ίδια κυβέρνηση. Βέβαια πιστεύω ότι το θέμα δεν είναι ακόμα, δεν έχει οριμάσει ακόμα και θα πρέπει να εμβαθύνουμε κάπως περισσότερο σε αυτή την ακρόαση και στη διακυβέρνηση. Τώρα, αυτά τα θέματα είναι θέματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε μια Τοματική κάπως διακυβέρνηση. Πρέπει να ε, βελτιώσουμε την κατάσταση, να είμαστε πιο επιθετικοί. Φυσικά θα πρέπει να κάνουμε στο τέλος μια σύνθεση όλων αυτών. Έχουμε κάποιες ε, εφαρμογές κλειδιά για την δημόσια διοίκηση να προσπαθήσουμε να τα αναπτύξουμε όλα αυτά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκείνες τις εφαρμογές επίσης που, έχουν, που διευκολύνουν την επαφή ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τη διοίκηση και αυτό το, το σημείο της διακυβέρνησης είναι κομβικό έτσι ώστε όλα αυτά τα εκατομμύρια ευρώ να επενδυθούν όσο γίνεται καλύτερα. Ε, κύριε Πρόεδρε, ήδη μίλησα αρκετή ώρα. Ε, θα ήθελα απλά να σας πω ότι εγώ και οι σκιώδεις εισηγητές. Θα θέλαμε ήδη να ευχαριστήσουμε τους εμπειρογνώμονες που θα μας μιλήσουν. Για μας είναι πολύ σαφής η κατάσταση. Είμαστε η πρώτη χώρα, η Πορτογαλία, όσον αφορά την ευρωπαϊκή κατάδειξη ε, ε, για την ε, Είμαστε στην πρώτη θέση της κατάταξης ε, όσον αφορά το διοικητικό μηχανισμό. Αν έπρεπε κανείς να μας δώσει ένα σημείο, ένα σημείο, ένα σημείο αναφοράς, είναι ο, η δόκτωρας που ε, σήμερα είναι ανάμεσα στους εμπειρογνώμονές μας. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την κυρία Λίζα Γιάκονσάρη που αντιπροσωπεύει σήμερα εδώ την ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας αγαπητοί συνάδελφοι και θα ήθελα να ακούσουμε τώρα τη δική σας γνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εφόσον όλοι ήδη φοράτε τα ακουστικά σας θα μιλήσω στα φιλανδικά. Την τελευταία έκδοση του περιοδικού Spiegel η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων μαζί με το μεγαλύτερο γερμανικό συνδικάτο είπαν, δήλωσαν ότι η ψηφιοποίηση θα είναι το θέμα κλειδί για φέτος. Και αυτό δείχνει απόλυτα σαφώς ότι η ψηφιοποίηση βρίσκεται στο επίκεντρο του θεματολογία μας. Φυσικά υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με την ψηφιοποίηση και οικονομικά μαθηματικά, αλγόριθμοι κτλ. Αλλά η ψηφιοποίηση είναι πολύ περισσότερο από αυτά. Πρόκειται για μια βιομηχανική επανάσταση στην ουσία που θα αλλάξει τα πάντα. Αλλάζει την εργασιακή ζωή, τις ανθρώπινες σχέσεις, τον πολιτισμό μας, αλλά και την κατανομή εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν να ανταποκριθεί σε αυτή την επανάσταση. Σε αυτή τη θητεία η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς είδε να διευρύνονται, μάλλον στην περασμένη, είδε να διευρύνονται οι αρμοδιότητές της και στην ψηφιοποίηση. Όσον αφορά δε, την προστασία του καταναλωτή, αυτή είναι τεραστία σημασία μέσα στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου και αυτό βέβαια αν κανείς δει ε, ποια είναι τα συμφέροντα των ε, επιχειρήσεων αλλά και των ε, ανθρώπων του κοινού ευρύτερα. Τώρα δυστυχώς υπάρχει αυτή η κοινή αρμοδιότητα ανάμεσα στην Ήτρε και στην ΙΜΚΟ και μας πήρε καιρό να ξεκαθαρίσουμε τα χωράφια μας, αλλά τώρα πρέπει να προχωρήσουμε πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, ελήφθη το ζήτημα των αρμοδιοτήτων και μπορούμε να αρχίσουμε την ε, ουσιαστική πια δουλειά εδώ εντό του Ευρωκοινοβουλίου. Τώρα, η δημοκρατική λήψη αποφάσεων σημαίνει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προφανώ ε, το Συμβούλιο επίση. και εμείς θα πρέπει να συνεργαστούμε, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε και με την ε, Επιτροπή η οποία πρέπει να προχωρήσει και εκείνη στις εργασίες της. Σύμφωνα με την πρόταση λοιπόν της Κομισιόν, το πρόγραμμα αυτό για την πρόθεση της διαλειτουργικότητας θα πρέπει να λειτουργήσει προς όφελος των καταναλωτών και των πολιτών και θα πρέπει πάνω απ' όλα να προωθήσει την συνεργασία εγώ από πλευρά τη ΣΥΜΚΟ θα ήθελα να πω ότι πρέπει να τονίσουμε κυρίως τον αντίκτυπο στους καταναλωτές αλλά και στις σχέσεις τους με τους διοικητικούς μηχανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στα θέματα που είναι ουσιαστικά για τους πολίτες. Δηλαδή, το θέμα του αλφαβητισμού στην ε, ε, ψηφιακή εποχή, γιατί υπάρχουν ε, άνθρωποι οι οποίοι είναι ε, γεννημένοι και εξοικειωμένοι στο ψηφιακά στην ψηφιακή εποχή, ενώ άλλοι που δεν έχουν σχέση πρέπει να καταρτιστούν. Οπότε θα πρέπει να βρούμε από κοινού την προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ξέρουμε πως η Επιτροπή σας, ΣΥΜΚΟ, συμμετέχει πλήρως στην έκθεση επί τη βάση του κανόνα 54 και μπορείτε με ουσιαστικό τρόπο να παρέμβετε στα αποτελέσματα ε, και να επηρεάσετε τη γνωμοδότησή μας και την έκθεσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την εισήγησή σας. Τώρα έχουμε την κυρία Γκέρτρου Δίνκεσταντ που είναι διευθύντρια του, ε, του τμήματος ε, ψηφιακέ λύσεις για τις επιχειρήσεις και θα ακούσουμε επίσης την κυρία Μαργαρίδα Βεκασής που είναι τμήματάρχης ε, του τμήματος ε, των διαλειτουργικών λύσεων για ε, την Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση. Προέρχεστε και οι δύο από την Γενική Διεύθυνση Digit της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω τώρα με ποια σειρά θέλετε να πάρετε το λόγο. Δυστυχώς. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο από 15 λεπτά και για τους, τις δυο σας. Ωραία, τότε θα σας κόψω 10 λεπτά. Άντε τώρα το είπα 15 λεπτά, εντάξει, εντάξει. Άμα μιλήσετε μόνο εσεί. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να τηρήσω τα 10 λεπτά μου έτσι κι αλλιώ, γιατί συνεργαζόμαστε πολύ στενά στην Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, uh, Ευχαριστώ και τα μέλη του Κοινοβουλίου. Είναι τιμή για μας να βρισκόμαστε εδώ. Με μεγάλη χαρά ακούσαμε ε, ότι θέλετε ε, να ακούσετε τη συνεισφορά μας και εμείς ε, προσβλέπουμε και επενδύουμε πάρα πολύ στη δική σας πρόταση και συνεισφορά για την επόμενη εργασία μας. Να πω όμως για την πρότασή μας πρώτα λίγα λόγια. Ποιο είναι το πολιτικό πλαίσιο. Έχουν και διαφάνειες, δεν θα μπορέσετε να τα δείτε όλα σε λεπτομέρειες. Ε, θα σας εξηγήσω εγώ τι γίνεται. Ο δημόσιος τομέας είναι βασικός ε, φορέας στην ευρωπαϊκή οικονομία και είναι ένα τμήμα της λύσης στην ε, χρηματοοικονομική κρίση. Το μισό δημόσιο ΕΠ, στο μισό ΕΠ, ε, στην Ευρώπη παράγεται από το δημόσιο τομέα, ο οποίος απασχολεί το 25% των εργαζομένων. 19% είναι οι δημόσιες συμβάσεις του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε βήμα προς τις ε, ηλεκτρονικές προκηρύξεις και διαγωνισμούς ε, θα σημαίνει τεράστιες οικονομίες για τα κράτη-μέλη κοινοτική αρμοδιότητα ε, στο δημόσιο τομέα δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ε, υπάρχουν ε, αρκετοί τομείς που είτε έμεσα είτε άμεσα επηρεάζουν αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα θα μπορούσα να αναφέρω η στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ψηφιακή ενιαγορά, αγορά, το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη που ήδη ακούστηκε και οι αιτήσει εκθέσεις για την ανάπτυξη, το ευρωπαϊκό εξάμεινο και ο εξυγχρονισμός ε, των ευρωπαϊκών δημοσίων διοικήσεων. Και ε, όλο και περισσότερο ζητούμε από το δημόσιο τομέα, από τις διοικήσεις να κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους. Για ποιο λόγο χρειάζεται ε, διαλειτουργικότητα. Τι σημαίνει αυτό. Είναι πολύ εντυπωσιακός ο όρος και πολύ ισχυρός. Θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο αποδοτικοί. Για να γίνει αυτό πρέπει οι μέθοδοι εργασίας μας στη δημόσια διοίκηση να ε, προσαρμοστούν, να εξυγχρονιστούν. Ποιες είναι αυτές οι αρχές. Ε, once only λέγεται στα ε, αγγλικά αυτό, δηλαδή μία φορά δίνεις τα στοιχεία σου είτε είσαι πολίτης είτε εταιρεία στη δημόσια διοίκηση και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και άλλες υπηρεσίες. Έχουμε τις λεγόμενες μόνο απευθυντικές θηρίδες που πας μόνο σε έναν άνθρωπο και απευθύνεσαι, one stop shop. Και να είναι ο κανόνας ε, το ηλεκτρονικό και το χαρτί να είναι εξαίρεση και να έχουμε λιγότερη διαπροσωπική επαφή με που τα πάντα ηλεκτρονικά αν γίνεται. Και ε, να συνδυάζονται τα στοιχεία σε διάφορες υπηρεσίες, να υπάρχει διάβγεια και διαφάνεια παντού στο δημόσιο τομέα, στις συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα για τις υπηρεσίες και ε, θα είναι ανοιχτά και στην πρόσβαση για το κοινό και για τις επιχειρήσεις. Να δημιουργούνται νέες υπηρεσίες λοιπόν ε, με διαφάνεια. Για να τα κάνουν όλα αυτά όμως χρειάζεται αλλαγή νοοτροπία στη δημόσια και συνεργασία, συνέργεια μεταξύ των διαφόρων υπουργείων και υπηρεσιών. Να ε, μην είναι κλειδωμένα τα δεδομένα και περιχαρακωμένα, να είναι πιο απλή η διαδικασία και να πέσουν οι φραγμοί και τα εμπόδια ανάμεσα στα διάφορα υπουργεία. Παντού το βλέπουμε αυτό. Χρειάζεται απλούστευση στι μεγάλε μηχανέ, στι διοικητικέ και αυτό είναι κάτι το οποίο καταπολεμάμε και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έχετε υπόψη σα. Για τα πολιτικά θέματα, η διαλειτουργικότητα είναι όλο και πιο σημαντικά. Το βλέπουμε αυτό και στην Ένωση. Όλο και περισσότερο έχουμε διασύνδεση και διαλειτουργικότητα σε πολλού τομεί. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από την Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επίτροποι και αντιπρόεδροι το έχουν ως μεγάλη προτεραιότητα αυτό και τα τρία τέταρτα των κρατών μελών επίσης. Οι ε, πρωθυπουργοί έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της διαλειτουργικότητας για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης τους. Έχει σημασία λοιπόν η διαλειτουργικότητα. Θα θέλαμε να σας δείξουμε ένα παράδειγμα τι οικονομίες μπορούν να γίνουν και πώς ε, μπορεί αυτό να επηρεάσει την οικονομία μας. Δεν βλέπετε τις λεπτομέρειες στη διαφάνεια γιατί είναι μικρά τα γράμματα εδώ και οι πίνακες. Η μελέτη αναρωτιέται εάν η διαλειτουργικότητα είναι κλειδί, όσο περισσότερο είναι διασυνδεδεμένα τα Υπουργεία και οι υπηρεσίες μεταξύ τους, τόσο λιγότερο χρόνο χρειάζεται ο πολίτης ε, να ε, σπαταλάει για να διεκπαιρέουν τις δουλειές του, χρόνο που θα τον αφιερώσει στην πραγματική οικονομία και στις δραστηριότητε του για να παράγει περισσότερα. Είναι παραγωγή του ΕΠ η ωραία εδώ, ε, ο δείκτης με τον οποίο μετράμε αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, αν έχουν 10 συναλλαγές διαπροσωπικές στο δημόσιο και κάθε συναλλαγή χρειάζεται μισή ώρα, οι απώλειες του ΑΕΠ στο Βέλγιο θα ήταν 2,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία 12,8 δισεκατομμύρια. Ε, ε, αυτά είναι πολλά λεφτά για να τα παραμελούμε έτσι και κάτι πρέπει να γίνει. Ε, ποιες είναι λοιπόν οι προκλήσεις, γιατί δεν το έχουμε ήδη καταφέρει αυτό. Αν είναι τόσο σημαντική η διαλειτουργικότητα και έχουμε ήδη κάνει τόσα πολλά. Παράδειγμα, η Σουηδία, που είναι η χώρα που γνωρίζω καλύτερα από τις υπόλοιπες είναι μέσα στις 10 πρώτες ε, ε, στην ε, χρήση του διαδικτύου, 93% των οικοκυριών. Και οι πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, τα άτομα δηλαδή, για τις συναλλαγές με το δημόσιο είναι 72%, μεγάλη εκτόση. Και ακόμα περισσότερο ε, είναι η απάντηση που δίνει το δημόσιο ηλεκτρονικά στους πολίτες, το 46%. Δηλαδή δεν αρκεί να έχει την υποδομή ως λύση, ούτε να έχεις την ψηφιακή διασύνδεση. Πρέπει να υπάρχει ουσιαστική διασύνδεση, αλλιώς ε, αλλιώς έχουμε κάθετη οργάνωση και όχι οριζόντια. Είναι βασικό αυτό. Δεν αρκεί λοιπόν η υποδομή, πρέπει να υπάρχει διασύνδεση οριζόντια εγκάρσια μεταξύ των υπηρεσιών. Έχουμε το πρόγραμμα αυτό ε, ε, ε ίσα στο τετράγωνο. Η λειτουργικότητα είναι μια προτεραιότητά μας εδώ και καιρό, αλλά μετά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε διαπιστώσαμε ότι πρέπει να γίνουν και περισσότερα. Να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία του παρελθόντος, να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή και τι σημαίνει αυτό. Έχουμε ένα πρόγραμμα με ένα μοναδικό στόχο, ενιαίο. Όπως και το προηγούμενο πρόγραμμα έχει στόχο να διευκολύνει την αποτελεσματική και αποδοτική ηλεκτρονική ε, επικοινωνία διασυνοριακά και διακλαδικά μεταξύ των ευρωπαϊκών δημοσίων διοικήσεων και των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ε, συμμετείχαν στα προηγούμενα προγράμματα αλλά σιωπηρά. Τώρα γίνεται ρητή αναφορά. Δείχνει λοιπόν το πρόγραμμα ότι υποστηρίζονται οι ανταλλαγές μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων που είναι οι άμεσοι ε, αποδέκτες αλλά και με τους εμέσους ε, δικαιούχους ας πούμε, οι υποφελούμενους που είναι οι πολίτες και επιχειρήσεις. Το πεδίο εφαρμογή έχει ενισχυθεί σε σχέση με το τρέχον πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα, όπως και προκάτοχος, θα εντοπίσει, θα δημιουργήσει και θα λειτουργεί τέτοιες λύσεις με ε, απεριόριστη χρήση και πρόσβαση σε άλλους θεσμούς ευρωπαϊκούς, τοπικούς, περιφερειακούς και λοιπά, σε κράτη-μέλη για να υποστηρίζεται η εφαρμογή και υλοποίηση των κοινοτικών πολιτικών, να εδρεωθεί, να προωθηθεί ε, το σημερινό πρόγραμμα και να επεκταθεί ε, και να ε, είναι και καταλήτης, να υποάζει λύσεις ας πούμε αυτό το πρόγραμμα για να μπορούν να ε, χρησιμοποιούμε την διευκόλυνση διασυνδέοντας την Ευρώπη ή άλλα μέσα για να φτάνουν όλα αυτά τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ενίος στόχος του προγράμματος υποστηρίζεται και από κάποιους λειτουργικούς στόχους που ονομάζονται προγραμματικές ε, ε, δραστηριότητες. Μπορούμε να το δούμε αυτό στο πρόγραμμα. Διατήρηση και χρησιμοποίηση των υφιστάμενων δομών διαλειτουργικότητας όπως ισχύουν σήμερα στο ΆΙΖΑ. Ε, η ανάπτυξη και επαναχρησιμοποίηση νέων δυνατοτήτων και νέων λύσεων διαλειτουργικότητας που υπάρχει και πάλι στο ΙΖΑ. Εκτίμηση πόσο θα επηρεάσει η τεχνολογία της πληροφορικής, την προτινόμενη κείμενη κοινοτική νομοθεσία για τα νέα μέτρα. Και πάλι αυτό υπάρχει στο πρόγραμμα ΕΙΖΑ. Ο εντοπισμός κάποιων νομοθετικών ελλημάτων ή κενών που εμποδίζουν την διαλειτουργικότητα. Και εδώ έρχομαι στο μέλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε καινούριο και τι βοηθάει. Το ΕΙΡΑ, το πρόγραμμα και το EIQ ε, ε, ΚΑΡΤ. Θα πρέπει να χαρτογραφηθούν οι λύσεις, να δημιουργηθεί, να συντηρηθεί και να επεκταθεί και αυτό το πρόγραμμα. Να δούμε ποιες είναι οι κοινέ προδιαγραφές και οι ειδικέ ρυθμίσεις και επίσης ανάπτυξη, ε, δρέωση και διεύρυνση νέων προτύπων και δομών. Ένας μηχανισμός που θα μπορεί να μετράει και να ποσοτικοποιεί τις λύσεις αυτές και αυτό πάλι καινούριο είναι. Και τώρα πώς μπορούμε αυτά να τα κάνουμε πράξη, αυτά που λείπουν εφόσον τα έχουμε εντοπίσει. Πώς ελέγχουμε λοιπόν και αξιολογούμε το πρόγραμμα αυτό. Όπως και τα προηγούμενα προγράμματα ε, είναι συνεχής η παρακολούθηση και τα αποτελέσματα ε, θα δημοσιεύονται επιγραμμικά ή θα είναι εύκολο κανείς να τα παρακολουθήσει. Θα υπάρξει μια διάμεση και μια τελική αξιολόγηση που θα διαβαστεί στο Κοινοβούλιο Υπάρχουν δείκτες που πρέπει να ε, μετρούν ε, την απόδοση του προγράμματος. Και έχουμε και μία πλήρη λίστα, ένα κατάλογο εξαντλητικό ε, δικτών, αλλά υπάρχουν και κάποιοι βασικοί καταλήτες ή διευκολυντές, αν θέλετε, για να πάρει μπρος το πρόγραμμα. Και θα πρέπει να είναι μετρημένο και μετρήσιμο το αποτέλεσμα και ο θετικός αντίκτυπος. Ε, ε, αυτά μας είναι ιδιαίτερα προσφυλή τα θέματα και πιέζουμε πάρα πολύ. Η διάρκεια είναι πενταετής, 2016 μέχρι 2020 και εντάσσεται πλήρως στο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο προπολογισμό είναι 131 εκατομμύρια, είναι πάνω κάτω το ίδιο με σήμερα, απλώς έχει μοιραστεί στα διάφορα χρόνια, 26 ε, ευρώ το χρόνο δηλαδή, για την πενταετία και το τελευταίο slide εδώ, η τελευταία διαφάνεια, συνοψίζει κάπως και τονίζει τα σημαντικά για μας θέματα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο ε, συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων Υπουργείων και Αρχών. Θα πρέπει τα αποτελέσματά μας να ε, διαδίδονται, να μην υπάρχει επικάλυψη και διπλό δηλαδή, ένα σαφές πλαίσιο για να αναπτύξουμε αυτές τις υπηρεσίες και τις λύσεις που να είναι ενίο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντα να έχουμε στο μυαλό μας την ευρύτερη εικόνα. Πού θέλουμε να πάμε και πώς θα φτάσουμε εκεί και τι θέλουμε να πετύχουμε, ποιος είναι ο στόχος μας. Δηλαδή να έχουμε μια καθολική, μια ολιστική προσέγγιση, να μην κοιτάμε μόνο το αυστηρά τοπικό ας πούμε και θα πρέπει ε, να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα που μπορούν να βοηθήσουν προς την κατήστηση αυτή. Τέλος, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε τώρα νέους επιτρόπους και με μια νέα ευκαιρία. Γιατί τονίζει πάρα πολύ τη συνεργασία η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεταξύ των επιτρόπων αλλά και σε επίπεδο των υπηρεσιών. Και ξέρουμε και από τις επαφές που έχουμε με τον έξω κόσμο και με τα κράτη-μέλη ότι καμιά φορά τους οδηγούμε σε σύγχυση. Έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές προτεραιότητες και, και πρωτοβουλίες και ο έξω κόσμος δεν βλέπει εκ πρώτης όψεως ότι όλα αυτά είναι συντονισμένα και τα θεωρεί συγκεχημένα ή κατακαιρματισμένα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι συνδέουμε τις δυνάμεις μας και έχουμε κοινούς στόχους τους οποίους και μπορούμε να δείξουμε προς τα έξω. Ότι είμαστε συντονισμένοι, ότι είναι κατανοητή η προσπάθειά μας αυτή για να εξυγχρονίσουμε τελικά τη δημόσια διοίκηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακρηγόρησα παραπάνω, μίλησα πόσο όσο περίμενα, υπέθετα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική σας παρουσίαση. Θα περάσουμε αμέσως στις μελέτες. is special advisor. Ε, λοιπόν, έχουμε την σύμβουλο της Deloitte, την κυρία Αναμπέλα Πετρόζο, η οποία θα παρουσιάσει την πρώτη περίπτωση αυτή της Πορτογαλίας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας ε, τα όσα έχουμε κάνει στην στρατηγική διαλειτουργικότητας ε, της ε, Πορτογαλίας και να σας αναφέρω κάποια πράγματα για το πρόγραμμα Αιζα 2. Μαργαρίτα. Α, μπράβο, ευχαριστώ. Η πρώτη διαφάνεια είναι ο δικός χάρτης και σας δείχνει την στρατηγική της πορτογαλικής κυβέρνησης που ξεκίνησε το 1999 με αυτό το οποίο λέγαμε τα ΚΕΠ τότε και δεν σταμάτησε έκτοτε εκεί πέρα λοιπόν στρατηγική αυτή έπαιζε σημαντικό ρόλο η πληροφορική και η διαλειτουργικότητα που έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να βάλει την ε, Πορτογαλία στη νέα εποχή και είχαμε την ευκαιρία να διδαχτούμε από άλλα κράτη-μέλη και να ευθυγραμμίσουμε την στρατηγική μας και να πω πως η ευκαιρία ε, αυτή του να μοιραστούν τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έτσι αυτό μου επιτρέπει στην περίπτωση, την... μας επέτρεψε στην περίπτωση της Πορτογαλίας να κάνουμε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ε, είχαμε παραδείγματος χάρη ε, συναδέλφους από το Βέλγιο που μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να μην κάνουμε λάθη. Οπότε το να κάθονται τα ίδια τα κράτη-μέλη στο ίδιο τραπέζι και να μοιράζονται ιδέες ή και λάθη μας έδωσε την ευκαιρία να βελτιωθούμε, οπότε θέλω να ευχαριστήσω τους Βέλγους ε, συναδέλφους ε, στους οποίους είμαι ευγνώμων. Δεύτερον, να αναφερθώ στην ε, επιτυχία μας στην ε, ιστορία, γιατί αν δεν σας δώσω κάποια πρακτικά παραδείγματα δεν θα μπορέσετε να αντιληφθείτε την δυσκολία του να έχουμε, να κάνουμε τα διάφορα βήματα, τα τεχνικά, τα οργανωτικά. Κοιτάξτε, η επιτυχία μας είχε μία πρακτική πλευρά που πρέπει να αντιληφθείτε γιατί αλλιώς δεν θα καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι να λειτουργήσουν τα διάφορα τεχνικά, σημασιολογικά και νομικά ζητήματα. Όλοι οι Πορτογάλοι απέκτησαν την ηλεκτρονική ταυτότητα. Γιατί? Γιατί είχε μία ιδιαιτερότητα που προκύπτει από το Σύνταγμά μας, που απαγορεύει να υπάρχει ένας φάκελος με όλες τις πληροφορίες για έναν πολίτη. Και βεβαίως ε, η πρόκληση αυτή μας έκανε να χρησιμοποιήσουμε κάποια πορτογαλική δημιουργικότητα και να χρησιμοποιήσουμε την ε, διαλειτουργικότητα ε, για να καταφέρουμε κάτι το οποίο ήταν αδύνατο. Να έχουμε μία κάρτα και ανεξάρτητα συστήματα πληροφοριών. Και έτσι ευθυγραμμίσαμε το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, τελικά, όχι, ο μεγαλύτερος αγώνας αφορούσε ακριβώς τις λέξεις ε, και την κάλυψη. Οπότε μετά από κάποιους αρχικούς περιορισμούς ε, έχουμε επιτύχει και τώρα έχουμε πάνω από 9 εκατομμύρια ταυτότητες που έχουμε παραδώσει και από το 2007 δεν έχει σταματήσει καθόλου ε, η διαλειτουργικότητα. Κάτι το οποίο μας δείχνει πως είναι δυνατόν να βελτιώνουμε την κατάσταση όμως πραγματικά υποφέραμε για να αποκτήσουμε αυτή την εμπειρία. Κάποιες από αυτές τις εμπειρίες θα μοιραστώ μαζί σας σήμερα γιατί υπάρχουν και κάποιες ομοιότητες με το ΆΙΖΑ. Το πρώτο μάθημα ήταν ότι έπρεπε να αλλάξουμε νοοτροπία. Να υπάρχει ευελιξία και να μην θεωρούμε ποτέ δεδομένο πως ό,τι θεωρούμε εμείς καλύτερο είναι αυτό το οποίο θέλουν οι άλλοι. Όταν ήμουν με τους συναδέλφους ήταν σαν τη συνάντηση με τα κράτη-μέλη. Ο καθένας ήταν ε, ξεχωριστός και είχαν δίκιο ναι, είχαν δίκιο, ήταν μοναδική, αλλά από τη δικιά μας την πλευρά έπρεπε να, αντιληφθούμε, να το αντιληφθούμε αυτό, να κάνουμε συμβιβασμούς, να υπάρχει ανθεκτικότητα και βεβαίως να μην υποχωρούμε ποτέ από τον στόχο μας. Το δεύτερο μάθημα ήταν να ε, είμαστε απλοί. Η πολυπλοκότητα του έργου ήταν τόσο μεγάλη που πραγματικά μας ξεπερνούσε ορισμένες φορές. Οπότε το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να τα σπάμε σε μικρά κομμάτια και να έχουμε κάποιες προτεραιότητες. Και τρίτον που προκύπτει από τα άλλα δύο, να ενσωματώσουμε τις ε, διαφορές και συνεχώς να ε, βελτιωνόμαστε. Και το τέταρτο και τελευταίο ήταν το εξής βεβαίως. Το νόημα των λέξεων όταν μιλάμε για αισθήματα προφορική, είναι απλό, μεταφράζουμε, συμφωνούμε, γίνεται κάτι τυποποιημένο και από εκεί και πέρα δεν το ξανασκεφτόμαστε. Με τους ανθρώπους όμως δυσκολεύουν τα πράγματα. Ακόμα και τώρα που σας μιλάω, καθένα από εσά θα καταλάβει κάτι διαφορετικό από τις λέξεις μου με βάση την δική σας ερμηνεία. Οπότε βασικές λέξεις όπως ευελιξία, απλότητα, το προτεραιότητα και όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίσει το ΆΙΖΑ 2. Επιτρέψατε μου λοιπόν να εκφράσω την άποψή μου για το νέο ΆΙΖΑ. Θα χρησιμοποιήσω εδώ πέρα τη λέξη του Αντιπρόεδρου της Κομισιόν γιατί συμφωνώ πλήρως. Έτη δουλειά στην διαλειτουργικότητα και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει τώρα να αποδείξουν την αξία τους και να ε, αποδώσουν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες για τους πολίτες και πιο φτηνά. Γι' αυτό ακριβώς, Μαργαρίτα, κοιτάω εγώ το πρόβλημα. Αυτό το Άιζα και το θεωρώ μια ευκαιρία και να υπάρχει και συνέχεια και ταυτόχρονα το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως ευκαιρία για να κάνουμε το μέσα και ταυτόχρονα να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σήμερα. Η ΆΙΖΑ ε, είναι ένα, το αποτέλεσμα 20 ετών εργασίας. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Μεγάλα δεδομένα, ανοιχτά δεδομένα, νέες λέξεις που δημιουργούν νέα διλήμματα. Ναι, αλλά πρέπει να τεθούν αυτά ενώπιον των κρατών μελών όλα αυτά τα εργαλεία, ή μεθοδολογίες πρέπει να τα χρησιμοποιούν μόνο οι κυβερνήσεις ή μπορούν να αποτελέσουν μια ευκαιρία να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Γιατί, κυρίες και κύριοι, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι σχεδόν τα ίδια με αυτά του παρελθόντος. Οι δυσκολίες παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών είναι μεγάλες τεράστιες καμιά φορά και πρέπει να επικεντρωθούμε σε νέους τρόπους διακυβέρνησης, σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα και να ανοίξουμε και την πόρτα σε άλλους ε, φορείς. Επίσης ε, βεβαίως το ζήτημα είναι η βιωσιμότητα. Τι θα γίνει με έργα τα οποία επέτυχαν όπως το STORK, το ES, οι ηλεκτρονικές προμήθειες κτλ. Όταν δεν θα είναι πλέον πιλωτικά. Ποιος θα τα εκμεταλλευτεί ή θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, την κεντρική χρήση τους για τα κράτη-μέλη. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζει η ΆΙΖΑ 2. Γι' αυτό ακριβώς εγώ θεωρώ πως είναι μια νέα αρχή. Ε, μια δυτή προσέγγιση χρειάζεται να δούμε δηλαδή τα θέματα αυτά και την ενοποίησή τους ως ένα μέσο ανοιχτής διακυβέρνησης και βέβαια να αποδώσουν αυτές οι επενδύσεις για όλους πολίτες και δημόσιες διοικήσεις και επιχειρήσεις. Και παρά τη Γενική Συμφωνία μεταξύ κρατών μελών για το ότι το ΆΙΖΑ 2 θα παραμείνει στην ε, διαλειτουργικότητα των κρατών μελών πρέπει να υπάρχει μια νέα στρατηγική και ακριβώς να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Εάν πραγματικά πιστεύουμε στην ανάγκη να ανοίξει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους πολίτες. Συμπερασματικά, η ΆΙΖΑ 2 είναι ένα καλό και απαραίτητο εργαλείο για την συνοχή και την ε, τεχνολογική τον τεχνολογικό διαμοιρασμό των δομένων μεταξύ των κρατών μελών. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζομαι. χρειαζόμαστε νέα έργα, όπως τα οποία θα λειτουργήσουν ως ε, ένα μέρος στο οποίο θα αναπτυχθούν νέες λύσεις ή θα είναι γέφυρα λύσεων για να χρησιμοποιήσουμε και ανοιχτές προδιαγραφές και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και το e-sense παρά τις επιφυλάξεις που έχω για το μέγεθός του το οποίο είναι μια ομπρέλα που καλύπτει πάρα πολλά έργα. Οπότε, συνοψίζοντας, χρειάζεται προληπτική δράση στην επικοινωνία με τα κράτη-μέλη, να εστιάζουμε να μην ξεχνάμε ποτέ πως ό,τι κάνουμε σε οποιαδήποτε γενική διεύθυνση, χώρα, τομέα, πρέπει να καταλήγει σε δημιουργία απασχόλησης, ποιότητα ζωής και ευτυχία για όλους τους Ευρωπαίους. Απλοποίηση. Να χρησιμοποιούμε τα τεχνολογικά εργαλεία για να απλοποιούμε τις ε, πολύπλοκες διασυνοριακές υπηρεσίες και να ξεκινήσουμε εντός ε, εισαγωγικών με τις πολύπλοκες τεχνολογικές διαδικασίες, αλλά βέβαια μην ξεχνάμε και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Και τέλος, διαφάνεια. Θεωρώ πως ε, μήκυο, ενώσεις, ε, κοινότητες, όλα αυτά είναι τμήμα της επιτυχίας. Η ΆΙΖΑ μπορεί να συνδέσει διαφορετικά τμήματα της κοινωνίας και να χρησιμοποιήσουμε τα όσα ήδη υπάρχουν για να τα χρησιμοποιήσουμε πιο κοντά στον κόσμο. Και έτσι η καινοτομία θα γίνει κοινωνική η οικονομία. Και έτσι, και με συγχωρείτε, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, έτσι θα εφαρμόσουμε τη γέφυρα μεταξύ ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ανοιχτή διακυβέρνηση. Πράγματι λοιπόν είναι δυνατόν να συμβεί αλλαγή και μας περιμένει. Γιατί να μην πειραματιστούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα μας πείσατε ακόμη περισσότερο μετά τη δικιά σας ομιλία. Οπότε, ωραία τατά. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα, ο κύριος Ρωμαντομόφσκι έχει τον λόγο, υφυπουργός ε, της ε, ε, ψηφιοποίησης στην Πολωνία επίσης για 10 λεπτά. Παρακαλώ να ξεκινήσετε την παρουσίασή σας και από την άλλη θα ήθελα να σας παρακαλέσω παρακαλέσω τον αντιπρόεδρο τον Μύρος Λαβλάμσδορφ αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας να αναλάβει αυτό στην Προεδρία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Κάποιος, κάποιος πρέπει να είναι εδώ να πάει στιγμή. Δεν αφήνω εγώ την έδρα του Προέδρου μόνο της. Ευχαριστώ dziękuję bardzo, panie przewodniczący.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 Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε σήμερα για τη βιομηχανική επανάσταση, μια τεράστια αλλαγή που οφείλεται ε, στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Όλο ένα περισσότερο η κλάδη της οικονομίας αυτή τη στιγμή ε, ε, αναπτύσσονται και εκεί μπορεί κανείς να έχει ηγετική θέση αρκεί να μπορεί να χειριστεί την ψηφιακή τεχνολογία. Ο ρόλος του διοικητικού μηχανισμού θα ήταν να διευκολύνει την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και να μειώσει τα κόστη της ε, δημόσιας διοίκησης. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να γίνουν διάφορες δράσεις και θα ήθελα να σας δώσω με απλά παραδείγματα ποια προσέγγιση εμείς επιλέξαμε στην Πολωνία όταν ε, θελήσαμε να θέσουμε σε εφαρμογή την διαλειτουργικότητα. Αυτό καταρχήν ε, έχει να κάνει με την υπέρβαση των ψηφιακών φραγμών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα συνοριακά τις συνοριακές, ε, τους συνοριακούς φραγμούς αλλά και τις ε, καθημερινές επιχειρηματικές συναλλαγές. Ε, θα σημαίνει επίσης ότι πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να είναι διαθέσιμες και σε ψηφιακές πλατφόρμες. Κάτι ακόμα, διάθεση των δημοσίων δεδομένων. Τέλος, προσπάθεια για μείωση του κόστους του δημόσιου τομέα. φαίνεται το πιο σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα είναι να γίνουν δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασυνοριακό επίπεδο δηλαδή. Και ένα καλό παράδειγμα εδώ είναι η εφαρμογή του κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον ηλεκτρονικό και ταυτότητα και τις ε, σχετικές υπηρεσίες, EIDAS. E Κάθε κράτος πρέπει να εφαρμόσει αυτό το κανονισμό. Ο στόχος είναι να, ε, να εγγυηθούμε ε, την ε, ασφαλή ταυτοποίηση και από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός θα προσπαθήσουμε επίσης να βασιστούμε σε ένα από τα projects που κάναμε στο παρελθόν, δηλαδή αυτό το project που ονομάζεται STOCK. Εκεί δημιουργήσαμε κάποια πρότυπα, τα οποία μετά δοκιμάσαμε, που ελπίζω πως θα είναι χρήσιμα για την εξέβρεση λύσεων μέσα στο πλαίσιο του ε, κανονισμού EIDAS. Τώρα για να γίνουν ε, αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές σε διάφορους τομείς. Ένας εξ αυτών είναι η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, δηλαδή πρόκειται για διοικητική εργασία. Έπειτα νέες λύσεις θα πρέπει να βρεθούν γιατί έχουμε τώρα ολοκληρώσει την ηλεκτρονική σφραγίδα που σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστούν νέες λύσεις και βεβαίως οι ισχύουσες λύσεις αυτή τη στιγμή θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες προτάσεις. για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια λύση σε, όλες, σε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών στη διαδικασία εφαρμογής θα είναι βέβαια τα στάνταρ, τα πρότυπα αναφοράς, τα οποία έχουμε ήδη επιτύχει όταν μιλούσαμε για τα πρότυπα Isaac. Να σας εξηγήσω λοιπόν τι κάναμε στην Πολωνία. Το πιο Ε, το πρώτο που κάναμε ήταν να, εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες. Δηλαδή η πρόκληση ήταν η πρόσβαση στα στοιχεία των δημοσίων μητρών. Έχουμε πάνω από 600 τέτοια μητρώα στην Πολωνία που είναι προβολικά πολλά. Δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα είχε ένα σύστημα πια όπου θα υπήρχαν συγκεντρωμένα όλα αυτά τα στοιχεία. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, κάναμε μια ανάλυση που μας έδειξε πως αρκεί να έχει κανείς πρόσβαση σε 100 βασικά ε, δεδομένα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται σε διάφορα μητρώα, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει διάφο... όλες τις στοιχείες που αφορούν το... ένα συγκεκριμένο φορολογούμενο. Για παράδειγμα, και αποφασίσαμε έτσι να φτιάξουμε μια πλατφόρμα για όλα τα στοιχεία που θα αποτελείται από λίγα αλλά, αλλά πολύ σημαντικά μητρώα. Η νέα χρήση επίσης των δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Επίσης έχουμε το outsourcing, κατά κάποιο τρόπο αγοράζουμε στοιχεία πολλές φορές και τα πληρώνουμε με δημόσια χρήματα. Για να εξασφαλίσουμε λοιπόν ε, την ευέλτιστη χρήση των δεδομένων από τη στιγμή που τα έχουμε πληρώσει, θέλουμε αυτά να μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιηθούν από ΜΚΟ ή επιχειρήσεις Στην περίπτωση της ε, Πολωνίας και πάλι η βασική πρόκληση ήταν να δούμε πώς θα χειριζόμασταν τα στοιχεία που υπήρχαν. Ήταν μια νέα αυτή η πρόκληση και για να μπορέσουμε να το, την ξεπεράσουμε ήταν σημαντικό να συνεργαστούν διάφορα επίπεδα ε, και έπειτα θέλαμε να έχουμε μια ειδική νομοθεσία που σαφώς θα έλεγε και θα περιέγραφε όλους τους μεμονωμένους κανονισμούς για την εκνεοχρήση των δεδομένων. Επίσης φτιάξαμε ένα ειδικό πόρταλ, έχετε εδώ τη διεύθυνση, όπου μπορούσε κανείς να βρει όλα τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα από τη δημόσια διοίκηση. Διαλειτουργικότητα. Αυτό σημαίνει και κόστος. Να δούμε δηλαδή και να εξετάσουμε τις οικονομικές στοιχείες, έτσι ώστε ε, ό,τι είναι νέο να δούμε τι κόστος επιφέρει. Βασικός στόχος λοιπόν του project αυτού ήταν να εισαχθούν συγκεκριμένα πρότυπα θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε και σε ένα χαμηλότερο επίπεδο, δηλαδή με πολύ πρακτικά προϊόντα τεχνολογίας. Για παράδειγμα, στην Πολωνία υπάρχουν διάφοροι τομείς όπου αποφασίσαμε να εργαστούμε επί συστημάτων που μετά τα διαθέσαμε σε διάφορες μονάδες της δημόσιας διοίκησης, όπως π.χ. Ε, η δωρεάν ψηφιακή ε, υπογραφή για πολίτες και οργανισμούς. Το δημόσιο προφίλ όπως λέγεται. Έχουμε επίση ένα σύστημα για την αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων ανάμεσα στα διάφορες υπηρεσίες στην Πολωνία. Ε, είναι δωρεάν. Και έχουμε και ένα, μια συγκεκριμένη ροή εργασίας για τα ηλεκτρονικά έγγραφα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε γραφείο της στην Πολωνία, πάλι δωρεάν. Βασικά λοιπόν η διαλειτουργικότητα είναι μια περίπλοκη διαδικασία όταν κανείς ξεκινήσει να την εφαρμόσει. Πρέπει να τη διαχειριστεί σε διάφορα επίπεδα και γι' αυτό συχνά είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει για να προωθήσουμε αυτό το project και να θαρρύνουμε τον κόσμο να το χρησιμοποιήσει. Εισάγουμε κανονισμούς σε διάφορα επίπεδα στην Πολωνία, ε, όπως το soft law είναι οι συστάσεις, το πρώτο, το χαμηλότερο επίπεδο. Έπειτα έχουμε φτιάξει καταλόγους με ένα σύνολο καλύτερων πρακτικών, δηλαδή κάποιων αρχών που μετά τις προωθούμε οποτεδήποτε αναπτύσσονται νέα συστήματα τεχνολογίας, της πληροφορίας. Συστάσεις λοιπόν είναι το πρώτο επίπεδο, μετά έχουμε νομικούς μηχανισμούς που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του στρατηγικού προγράμματος που μας επιτρέπει να ε, ενσωματώσουμε τα μεμονωμένα προγράμματα σε ένα ευρύτερο σύστημα. Επόμενο επίπεδο, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την διαλειτουργικότητα. Εδώ ερχόμαστε στην οικονομική πτυχή, στη δημοσιονομική πτυχή. Έχουμε ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα που λέγεται Ψηφιακή Πολωνία. Mm. Και αγκαλιάζει όλα τα προγράμματα που σχετίζονται με την ψηφιακή ατζέντα, ευρυζωνικά δίκτυα, ε, συνειδητοποίηση, ενημέρωση για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ένα σωρό άλλα. Ένα από τα στοιχεία κλειδιά ή μάλλον τα κριτήρια ε, που θα πρέπει να επιτευχθούν ώστε να μπορέσουμε να έχουμε χρηματοδότηση, να μάλλον ο καθένας δεν μπορεί να έχει χρηματοδότηση, είναι ότι όντως στηρεί αυτές τις αρχές των οποίων στόχος είναι η πρόθεση της διαλειτουργικότητας. Αυτά λοιπόν και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε ε, Ντουμόφσκι. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Γνωρίζω κάπως την κατάσταση στη Πολωνία. Είμαστε γείτονες. Εγώ είμαι από την Τεχεία και γνωρίζω πως ε, Αυτό το γνωρίζω γιατί πολλές από τις εμπειρίες αυτές τις πολύ μπορούν να μεταφερθούν και να χρησιμοποιηθούν και στις γειτονικές χώρες. Αυτή η εισήγηση δείχνει την σημασία της αποκέντρωσης. Διότι σε μια τόσο μεγάλη χώρα είναι δύσκολο να κανείς να συγκεντρώσει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την διαλειτουργικότητα. Εγώ όταν με σπούδαζα την ιστορία του management, της διαχείρισης, θα πρέπει να πω ότι το πρώτο σχήμα το οποίο ακολούθησαν πολλοί άλλοι ειδικοί αργότερα ήταν ένα συγκεντρωτικό σύστημα διαχείρισης των Αμερικανικών σιδηροδρόμων. Αυτό μελετούσαμε τότε. Και μετά φάνηκε πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάντοτε αυτό. Η πρόοδος μέσω των ε, τεχνολογιών της πληροφορίας μας επέτρεψαν να αποκεντρώσουμε τη δημοσιοδίκηση και ελπίζω πως αυτή η αποκέντρωση θα συνεχιστεί και στο μέλλον γιατί αυτό είναι ο τρόπος για να είναι πιο αποδοτικό το σύστημα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζωγίνιο, που είναι εδώ. Ε, είναι άνθρωπος πάρα πολύ υπεύθυνο γιατί πέμπτη απόγευμα τώρα τέτοιες ώρες ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του. Ο συγητής έχετε μέσα στο λόγο κύριε Ζωρίνιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έκανα την ε, αρχική εισήγηση. Οι παρουσιάσεις που έγιναν αντιστοιχούν ε, άμεσα με τις προκλήσεις που έχουμε θέσει, έχουμε ορίσει, είναι η πραγματικότητα ότι τη σήμερα ημέρα και επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να το αναφέρω αυτό, ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το σύστημα διαχείρισης των Αμερικανικών σιδηροδρόμων και ακριβώς αυτό έχουμε ανάγκη να αποκεντρώσουμε και να, αλλά και να μιλήσουμε κοινή γλώσσα. Ταυτόχρονα τα νέα τεχνολογικά εργαλεία αλλά και η διαλειτουργικότητα είναι αυτά που μας επιτρέπουν να λάβουμε αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά να μπορέσουμε κιόλας να ομοδοποιήσουμε, όπως ε, είδαμε και από το παράδειγμα, το της Πολωνίας ή όπως είδαμε και από την Πορτογαλία και εδώ θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά ε, η ε, δόκτωρα Αναμπέλα Πεδρόζο έχει πια πάρει σύνταξη από το δημόσιο τομέα και είναι σύμβουλος μιας επιχείρησης στην οποία αναφέρθηκε αλλά η δοκτωρα σαναμπελα πεδροζο εχει πια παρει συνταξη απο το δημοσιο τομεα και ειναι συμβουλος μιας επιχειρησης στην οποια αναφερθηκε αλλα η δουλεια που έκανε έγινε ενώ ε, διατελούσε πρόεδρος του πορτογαλικού οργανισμού εναρμόνισης δηλαδή ε, ήταν ε, υψηλή αξιωματούχος του Πορτογαλικού κράτους και μπόρεσε να ε, μπόρεσε να τα ομαδοποιήσει, να ομαδοποιήσουμε όχι μια ενιαία μόνο κάρτα ε, ταυτότητα, αλλά μπορέσαμε έτσι να μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε όλα του τα στοιχεία, ανεξάρτητα από ποια δημόσια υπηρεσία αυτά είναι κατατεθειμένα ή ε, αποθηκευμένα. Γι' αυτό ήθελα να πω ότι αυτό το πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και με τους πολίτες. Δηλαδή διαλειτουργικότητα όχι μόνο ανάμεσα στις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, αλλά και με τους πολίτες. Οι άτυπε συζητήσει που έκαναμε με τον Πίτροπο και με, με την Επιτροπή, μάλλον και με του υπόλοιπου και ηγητή, ε, μα οδήγησαν στην σημερινή αυτή ακρόαση που, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ καλύτερη από ό,τι αρχική. Και αυτό είναι που και μα ενδιαφέρει. Δεν μα ενδιαφέρει ποιο κάνει τι, αλλά να μπορέσουμε να βρούμε κοινέ λύσει και να συγκλίνουμε προς τι ίδιε κοινέ λύσει. Η κυρία Ινστιτ είπε ότι η συνεργασία των εταιριών και των πολιτών εννοείται σε όλα αυτά. Δεν πρέπει πια να εννοείται, πρέπει να είναι σαφής ρητή. Γιατί όπως είπε η Αναμπέλα, ποτέ δεν θεωρήσαμε σίγουρο είναι αυτονόητο αυτό που ήθελαν οι άλλοι. Έπρεπε ε, να καλέσουμε τον κόσμο να μας πει τι επιθυμεί και αυτό είναι ένα βήμα που κάνει τη διαφορά. Και νομίζω και εμείς αυτό το βήμα θα πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή τη σύνοψη στην ιστορία. Οι Πορτογάλοι ανακάλυψαν για μας τους ωκεανούς. Ίσως ο κύριος Σορίνιο τώρα ανακαλύψει για μας ε, τα μυστικά της διαλειτουργικότητας. Κοιτάξτε, στο παρελθόν μπορεί να ανακάλυψε ε, τις, ε, τους ωκεανούς. Τώρα είναι η μόνη χώρα που διαχειρίζεται και τα νέφη, το cloud. Η κυρία ε, Γιάκο είναι επόμενη ομιλήτρια, η οποία είναι και σκιώδης εισηγήτρια. Μάλλον, συγγνώμη, συντάκτρια γνωμοδότηση της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους. Ήταν συναρπαστικές οι παρουσιάσεις. Ειδικά η περίπτωση της Πορτογαλίας εξαιρετική και χάρηκα πάρα πολύ που την άκουσα. Με, δηλαδή έχετε μέχρι και ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ε, μπράβο σας. και να πω και στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το ISA 2 είναι πάρα πολύ αφηρημένο, όσο ε, καταπληκτικούς στόχους και να έχει. Αλλά ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που θα πρέπει να γίνουν για την ε, ψηφιακή υποδομή και πέρα από την υποδομή. Χρειάζονται και τεχνολογικές αλλαγές καμιά φορά. Εσείς είστε ειδικοί, πώς θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε και να κάνετε κάποια πρόβλεψη πώς θα γίνουν όλα αυτά, πώς θα μεταφραστούν στην πράξη. Ο Ευρωπαίος πολίτης δεν είναι ενιαίος. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν δυσκολία ε, στο διάβασμα, δηλαδή είναι αναλφάβητοι. Μπορεί να είναι πολύ μικρό το ποσοστό, αλλά υπάρχουν. Να μην δημιουργήσουμε χάσματα τώρα και ρήγματα στον πληθυσμό δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ψηφιακά ορφανά, δηλαδή ανθρώπου που να είναι αποκλεισμένα από τη διαδικασία αυτή, γιατί δεν έχουν υπολογιστεί καν ή δεν ξέρουν ε, γραφή και ανάγνωση και δεν μπορούν ε, να απευθυνθούν ας πούμε σε μια κλινική, σε ένα κέντρο υγείας ε, ή σε μια δημόσια υπηρεσία για κάποιες βασικές υπηρεσίες. Αν όλα αυτά έχουν γίνει ψηφιακά, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα αποκλειστούν. Για παράδειγμα, στην Εστονία ε, διοργανώνουν μαθήματα για ε, ενταξιούχους και ηλικιωμένους για το διαδίκτυο και παρά το γεγονός ότι τους εκπαιδεύουν, οι άνθρωποι δεν έχουν υπολογιστή. Μπορεί να ξέρουν να το χειρίζονται, αλλά πρέπει να το βρουν. Πώς θα φτάσουμε πιο κοντά στους πολίτες, δηλαδή αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ. The next speaker ε, Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μπονέ, ευχαριστώ την κυρία Γιακονσάρη. Είναι πραγματικά ε, πρόβλημα αυτό ε, του αναλφαβητισμού σε πολλές περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήταν πολύ υψηλό και στο νότο της Ευρώπης. Αυτές οι δημοκρατικές πώς να το πω, εξελίξεις θα μας βοηθήσουν και η τεχνολογία να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν. Επόμενο ομιλητή, ο κύριο Μπόνι, που είναι σκιώδη εισηγητή από πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπόθηκαν όλα ήδη. Δύσκολο να μιλήσει μετά από όλου αυτού του ομιλητέ και να πει κάτι καινούριο. Θέλω όμω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και την κυρία Πετρόσο και τον κύριο Δημόφσκι που μας παρουσίασαν τις περιπτώσεις αυτές οι ειδικές των κρατών μελών και πώς μπορεί κανείς να διαχειρίζεται στην πράξη τη διελτουργικότητα. Θέτοντας προτεραιότητες, όπως έβαλε η Πολωνία, αλλά και με πολλές νέες λύσεις και στην Πορτογαλία. Έχει σημασία να καταλάβουμε στην Πορτογαλία με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες εννοώ. Ε, και το είπαν και οι ίδιοι. Ε, ε, η ανοιχτή διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Διαφανής δηλαδή με διάβγεια. Ήταν εξαιρετική η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί εμείς συζητάμε τώρα για το διακανονισμό και τα προγράμματα, λες και ήταν κάποιο είδους τεχνική λύση. Δεν ισχύει αυτό. Και σήμερα χάρη και στην ακρόαση αυτή, καταλαβαίνουμε καλύτερα ότι δεν είναι μόνο τεχνικό πρόβλημα αυτό, η τεχνική λύση, η τεχνολογική. Είναι ουσιαστικό για την ε, ενιαία ψηφιακή αγορά ως βάση και επίσης είναι ε, κομβικό για ένα νέο μοντέλο δημοκρατίας και ανοιχτής ε, διαφανούς διακυβέρνησης. Είναι πολύ χρήσιμο λοιπόν και καλά θα έκαναν ε, και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενέχονται περισσότερο σε αυτή την προσπάθεια και να διαδίδουν και τη γνώση για το πρόγραμμα αυτό στις χώρες μας. Μία ερώτηση έχω μόνο, την εξή, δύο. Πρώτον, τα προγράμματα ΆΙΣΑ και οι δράσεις πώς ανταποκρίνονται στην πράξη σε σχέση με τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν στην Πολωνία, Πορτογαλία και σε άλλα κράτη-μέλη. Και η δεύτερη ερώτηση, τι είδους νομοθετικό κενό διαπιστώνεται όταν υπάρχει ανάγκη να περάσουμε σε πιο βαθιά διαλειτουργικότητα, γιατί το ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι υπάρχει νομοθετικό κενό κάπου ή έλλειμμα ή χάσμα Καλό θα είναι λοιπόν εκ των προτέρων και όσο γίνεται πιο νωρί να εντοπιστεί αυτό και καλώς ορίζουμε τη δέσμη των μέτρων. Αλλά προβλέπετε και νομοθετικές αλλαγές πριν εφαρμοστεί. Γιατί, πώς να το πω, θα είναι τμήμα του ε, πακέτου για την ενιαία ψηφιακή αγορά που θα μας παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο. Ευχαριστώ κύριε Μπόνη. Τώρα, φιλελεύθεροι και δημοκράτες, ο κύριος Τόιρερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και τις πτυχές ε, και πληροφορίες που εκθέσατε. Όταν μιλάμε για την διαλειτουργικότητα βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές πτυχές. Αφενός έχουμε το ότι πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη ε, τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και το εάν ε, οι δημόσιες διοικήσεις στα κράτη-μέλη έχουν περάσει στην ψηφιακή εποχή, οπότε το θέμα είναι ποια είναι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αποστολή της βεβαίως είναι όταν μιλάμε για διασυνοριακές ε, ε, για διασυνοριακή λειτουργικότητα εντός Ένωσης. Και βεβαίω πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ε, εκ των προτέρων δεν σημαίνει πως τα πάντα είναι αυτομάτως αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το σκεφτούμε θα δούμε πως σε μια ανοιχτή ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να δημιουργηθούν ε, συνθήκες πλαίσιο γιατί χωρίς αυτές δεν γίνεται. Και βεβαίως εμείς ε, συνεννοηθήκαμε εδώ πέρα ε, πως η Επιτροπή Βιομηχανίας θα ασχοληθεί με τα θέματα της τεχνολογίας και όχι της προστασίας δεδομένων. Αλλά είναι πολιτική σχιζοφρένεια αυτό βεβαίως, γιατί ξέρω πάρα πολλούς πολίτες οι οποίοι είναι ε, οπωσδήποτε υπέρ της περαιτέρω ψηφιοποίησης ε, των διαδικασιών, αλλά και υπέρ της περισσότερης προστασίας των δεδομένων τους. Εάν δούμε το τι γίνεται στην Αμερικανική νομοθεσία, υπάρχουν ε, διασφαλίσεις για το ότι δεν επιτρέπεται ε, να αποθηκευτούν σε μαγνητικά μέσα εκτός είπα τα δεδομένα τους. Οπότε θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα αυτό προστασίας δεδομένων πανευρωπαϊκά θεωρώ εγώ. Γι' αυτό ακριβώς ε, ε, πρόκειται για ένα βασικό και αναπόσπαστο τμήμα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το ερώτημά μου τώρα. είναι τεχνικό όντως το ζήτημα του εάν μέσα από το Open Government θα βελτιώσουμε την κατάσταση ή είναι ρυθμιστικό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια διαδικασία πλαίσιο για να δώσουμε μία όθηση στην όλη κατάσταση. Θεωρώ λοιπόν πως ε, η Κομισιόν ε, είναι αρκετά επιφυλακτική ακόμα. Θα δούμε, αναμένω και τη συζήτηση με τα κράτη-μέλη λοιπόν. Ο πρόεδρος, ε, δεν ξέρω, μπορεί ακριβώ το πρόβλημα να είναι αυτή η ζώνη που αναφέρεται γιατί θα υπάρξει μια ψυχιακή επανάσταση. Πρέπει να το δούμε λοιπόν. Ο ναι. κύριος Μαραγκάλ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σήμερα, πολύ δε περισσότερο ακούγοντας τι διάφορες περιπτώσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εκπροσώπους, ε, Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με τους στόχους και όλα αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλές οι προοπτικές και ελπιδοφόρες. Αν με ρωτούσατε να σας πω τι περιμένω από το ίσα 2 είναι να μην υπάρξει ίσα 3. Να μην χρειαστεί δηλαδή να φτάσουμε σε ένα τρίτο πρόγραμμα. Γιατί θα έχουμε καταφέρει να εδραιώσουμε, να εγκαταστήσουμε έτσι το πρόγραμμα και το 2020 πια να είναι στην αιχμή του δόρατος και να είναι μια κανονικότητα, μια ομαλότητα, να μην χρειάζεται και ένα τρίτο πρόγραμμα. Ε, ούτε να φροντίζουμε γενικά να εφαρμόζεται σε κάθε χώρα, να είναι δεδομένο. Βεβαίως θα χρειάζεται διαχείριση ακόμα, θα πρέπει να έχουμε μια επαρκή βάση διαχείρισης, σύγκλησης των διαφορών, ε, βελτίωση, φυσική εξέλιξη κτλ. Αλλά να έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα, μια ομαλότητα, μια κοινή γλώσσα ε, Τη ψηφιακής χρήσης στην Ευρώπη, βέβαια πάντα με τις ιδιαιτερότητες του καθενός, ε, θεσμικές, εθνικές, ε, πολιτισμικές κτλ. Έλεγε η κυρία Πεντρόσο στην παρουσίασή της, keep simple, προσοχή στη σημειολογία και απλότητα. Θα προσπαθήσω τις επόμενες εβδομάδες και μήνες να ασχοληθώ με το θέμα αυτό και με μεγάλη χαρά θα το κάνω στο πλευρό του κυρίου Σωρίνιο. Θέλω να πω σύντομα τα εξή τέσσερα. Πρώτο, μπορεί να μην είναι στο σημερινό κείμενο, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν στόχοι σαφώς ορισμένοι και γενικοί και ειδικοί που να συμπληρώνονται από διάφορους παράγοντες με τον οδικό χάρτη αυτό το κρίσιμο για την ε, διαδικασία με ορόσημα περιοδικά ή ετήσια για να αξιολογούμε και τα μέσα αντικτύπου και τους στόχους που εκ των προτέρων έχουν οριστεί. Δεύτερον, το πρόγραμμα θα πρέπει να ορίσει συγκεκριμένες έννοιες, υπόθηκε. Θα πρέπει να κερδιθεί η σημασιολογική αυτή η μάχη. Να διευκρινίσουμε ποιες είναι οι προσδοκίες του καθενός και οι δυνατότητες του. Ρητά. Τρίτον, Ειλικρινά πιστεύω, το προτείνω, δεν ξέρω, στην αρχική παρουσίαση δεν το είδα, σήμερα κάπως καλύτερα ε, ακούστηκε αυτό. Θα πρέπει να επικεντρώνεται το πρόγραμμα στις γενικές συμφωνίες για ένα κοινό πλαίσιο. Κοινούς κανόνες παιχνιδιού, ας το πούμε. Και προδιαγραφές, πρότυπα και προαπαιτούμενα που θα πρέπει οι φυστάμενες λύσεις να συμπεριλαμβάνουν. Και πολύ περισσότερο από όλα αυτά πιστεύω ότι η συγκεκριμένη παραγωγή λύσεων, ειδικών ή γενικών, για όλες τις συναλλαγές ε, με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, ε, θα πρέπει να προσφέρεται αυτό το πλαίσιο. Η κυρία Αγγίστα τα εξήγησε σήμερα πολύ καλύτερα από την προηγούμενη φορά είχαμε ακούσει. Ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και αυτό που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσουμε την πρόσβαση των περιεχομένων στο διαδίκτυο, στο web. Για να καταλάβουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και ένα τέταρτο και τελευταίο, δεν το άκουσα πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα και να ε, ενσωματώνει ε, προηγούμενες επιτυχίες του προγράμματος αυτού του ίσα ή άλλων προγραμμάτων. Για παράδειγμα, Μιλάμε για πιλωτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας που τελικά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα e-sense. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλη τη δουλειά που έχει ήδη γίνει. Δηλαδή να απαιτούμε από τους αυτούς μας ένα στοιχειώδη συντονισμό για να αξιοποιούμε και να εκμεταλλευόμαστε το ε, βαθμολόγιο που ήδη υπάρχει. Δεν θα πρέπει να επανεφευρίσκουμε τον τροχό κάθε φορά. και επίσης να σπάσουν αυτά τα σιλό, αυτές οι κάθετες δομές, ε, ε, οι οργανικές σε διάφορες ε, διοικήσεις ή υπουργεία που δεν μας επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία τέτοιου είδους προγραμμάτων. Είμαι πεπισμένος ότι θα το επιτύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. And uh, the second part of our session, today's session, will be... Uh, Ευχαριστώ και το δεύτερο τμήμα της από μας ε, συνεδρίασης θα ξεκινήσει με τον Μπλάνκο Λόπες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του και για τις ε, πληροφορίες που μας προσέφερε μέσω αυτής της ακρόασης. Πιστεύω πως αυτή η εργασία εστίασε κυρίως ε, στην ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που, είναι, που, δίνει, που δίνει την έμφαση στις κοινωνικές πτυχές, στο πώς θα μπορέσουν δηλαδή οι δημόσιοι μηχανισμοί να ξεπεράσουν τις ψηφιακές δυσκολίες και πώς θα μπορέσουν να ξεπεράσουν όλα αυτά, τα, να, να μετατρέψουν μάλλον σε πράξη όλα αυτά που κρύβονται μέσα στις ε, κοινωνικές συνθήκες. Ε, αυτή λοιπόν την πιο κοινωνική πτυχή, εγώ θα υποβάλω κάποιες ε, τροπολογίες με αυτό το θέμα, αλλά θα ήθελα να θέσω και ένα θέμα στο οποίο αποδίδω τεράστια σημασία. Να γνωρίζω πως είναι σχεδόν μανία μου, δηλαδή η δημογραφική πρόκληση εκτός από την ε, μέσα μάλλον από την προπτική των δημοσίων ε, μηχανισμών. Εδώ η χρήση της τεχνολογίας, της πληροφορίας, η επικοινωνία, η διαλειτουργικότητα μπορούν και οφείλουν να παίξουν ε, ρόλο πολύ σημαντικό σε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και οι σχέσεις ανάμεσα στους διοικητικούς μηχανισμούς, στις επιχειρήσεις και τους πολίτες ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες περιστάσεις όπου βρίσκεται συγκεκριμένη εταιρεία ή πολίτης. Οι δημόσιοι μηχανισμοί θα πρέπει να συμβάλλουν στην υπέρβαση του φραγμού του ψηφιακού φράγματος, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου είναι πιο δύσκολο να γίνουν ε, επενδύσεις. Και γι' αυτό και εκτιμώ την προσπάθεια του εισηγητή για να εισάγει την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων στα θέματα της ιδιωτικής σφαίρας και της προστασίας των δεδομένων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο και Κάλλας. Κυρία Κάλλας, από την άλλη. Μάλιστα, ευχαριστώ. Έχω μια σειρά από να απευθύνω στους εκπροσώπους της Κομισιόν. Έχω μια δυσκολία να διακρίνω τι είναι νέο και τι προκύπτει από την ΆΙΣΑ. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι τα βασικά διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε από την εμπειρία της ε, ΆΙΣΑ και επίσης ποια είναι η αντιστοιχεία της κατανομής της χρηματοδότησης ανάμεσα στις διάφορες προτεραιότητες. Δηλαδή πώς αυτό έχει αλλάξει από την ε, ΆΙΣΑ. Ένα άλλο σύνολο ερωτήσεων αφορά τις σχέσεις με τα κράτη-μέλη η ΆΙΣΑ θα μπορέσει να στηρίξει τις περιφερειακές πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πανευρωπαϊκές λύσεις. Και ένα ζήτημα που έθιξε κυρίως η ενδιάμεση έκθεση είναι η συμμετοχή, η εμπλοκή μάλλον των κρατών μελών. Πώς αυτό θα ληφθεί υπόψη από την ΆΙΣΑ 2 και τι μπορούν να κάνουν καλύτερα τα κράτη-μέλη. Και έπειτα, μέθοδοι εργασίας. Πώς το πρόγραμμα ΙΣΑ 2 θα ε, συνδυαστεί με άλλα προγράμματα, πώς εντάσσεται στη νέα ιεραρχία της Κομισιόν και ποιος επίτροπος θα είναι υπεύθυνο. Πώς το ΙΣΑ θα επηρεάσει άλλες ε, υπηρεσίες και προγράμματα. Το ΆΙΖΑ 2 μπορεί να συνδυαστεί με προγράμματα που είναι επιλέξιμα για το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Ναι, τις απαντήσεις θα τις δώσουν οι εμπειρογνώμονες. Λοιπόν, σε αυτό το τμήμα τελευταίος ομιλητής είναι η κυρία Ντάλι από τους σοσιαλιστές. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ήθελα... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συγχαρώ τους, ε, τις εισηγήτρες γιατί κατάφεραν να αναπτερώσουν το ενδιαφέρον μας και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Μιλώ εξ ονόματος ε, των ε, σοσιαλδημοκρατών στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και Βεβαίω αυτό είναι σημαντικό το θέμα γιατί μιλάμε για τις ε, πληροφορίες για τους πολίτες αλλά μιλήσαμε και για την ε, ευτυχία. Και υπάρχουν τώρα δύο σημεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Κάτι το οποίο μας απασχολεί εμάς ε, στους σοσιαλδημοκράτες και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναρμόνιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και υπάρχουν διάφοροι κανόνες όσον αφορά τις υποχρεώσεις των κρατών μελών. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκληση μεταξύ των όσων ισχύουν στα διάφορα κράτη-μέλη και προφανώς μια τέτοια κατάσταση σημαίνει πως δεν θα έχουμε 100% διαλειτουργικότητα δεδομένου του ότι βασικό κομμάτι της ε, διαλειτουργικότητας είναι οι ίδιες προδιαγραφές και κριτήρια σε όλα τα κρατημέλη. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε επιγόντως. Γι' αυτό ζητάω την γρήγορη υιοθέτηση του πακέτου προστασίας προσωπικών δεδομένων γιατί έχει κολλήσει στο Συμβούλιο. Εδώ και καιρό το Κοινοβούλιο περιμένει για να διαπιστώσει πώς θα είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ίδιες προδιαγραφές και αυτό θα ωφελήσει τους πολίτες και το δημόσιο τομέα. Ένα άλλο, ένα άλλο τελευταίο θέμα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται βεβαίω με την ε, αρχική ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, αλλά η Κομισιόν θα πρέπει να καθορίσει πως οι εταιρείες οι οποίες ε, υποβάλλουν τις προτάσεις τους πρέπει να καθορίζουν το πώς αναφέρονται στην ε, προστασία δεδομένων. Αυτό ιδιαίτερα για οτιδήποτε αφορά τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ που αναφέρατε το θέμα αυτό. γιατί Βεβαίω ασχολούμαστε με την προστασία δεδομένων, αλλά δεν είχαμε αναφερθεί αρκετά. Τώρα λοιπόν, με την αδειά σα, θα διαβάσω αυτά τα οποία έχει να πει ο συνάδελφος από την η συνάδελφος, η Μαρίζα Ματίας και ο Δησηγήτρια, η οποία τελικά αλλά ίσως είναι καλύτερο να δώσουμε τον λόγο στους ειδικούς. Νομίζω το καλύτερο είναι αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Γκέρτρουντ Ίγκεστατ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα, θα παραχωρήσω τον ε, λόγο αμέσως στη Μαργαρίτα για να μας πει εκείνη. Κυρία Μπεκαζές. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Γερτρούδη, θα προσπαθήσουμε να δούμε κάποια από τα ζητήματα αυτά που έτεθησαν. Πρώτα απ' όλα. Η κυρία Γεκονσάρη έφυγε, αλλά να ξεκινήσω με την δικιά της ε, παρέμβαση. Το βασικό στόχος είναι να χτίσουμε τα θεμέλια, όπως είπε πριν ο κύριος ε, βουλευτής, και πάνω εκεί πέρα θα οικοδομήσουμε το σύστημα και θα βρούμε τις λύσεις ε, στις διάφορες διοικήσεις. Έχουμε λοιπόν, αν θέλετε, διάφορα κομμάτια, τούβλα, με τα οποία θα χτίσουμε τις διάφορες λύσεις. Να αναφέρω την πτυχή ε, που ακούστηκε και είναι σημαντική. και θα συνεχίσει να μας απασχολεί αν υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τους όρους, την ορολογία. Δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μεταξύ ε, διοικήσεων χωρίς να συμφωνήσουμε για την ορολογία. Και ορολογία διατομεακή γιατί οι άνθρωποι του ίδιου τομέα συνεννοούνται και καταλαβαίνουν τι εννοούν με τις λέξεις που χρησιμοποιούν αλλά όταν μιλάμε για άλλους τομείς δεν είναι τόσο απλό. Οπότε εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα του πόσο σημαντική είναι η δουλειά του προγράμματος ΆΙΖΑ. Να μπορέσουν δηλαδή διάφοροι φορείς να συμφωνήσουν στην ίδια ορολογία και έχουμε κάποιες επιτυχίες. με τα, την ορλογία που έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Δεν θέμε ορφανά και ψηφιακό χάσμα. Οι λύσεις, ε, τα πλαίσια τα οποία προτείνονται με την βοήθεια των κρατών μελών ε, από μόνα τους δεν συνεισφέρουν σε ένα ψηφιακό χάσμα προσφέρουν λύσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και κατά κανέναν τρόπο δεν αποτρέπουν τη λήψη μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψη τους ανθρώπους που δεν είναι συνδεδεμένοι. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια αντίφαση. Μπορούμε να έχουμε κάποιες λύσεις για την πλειοψηφία του πληθυσμού και ταυτόχρονα να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες αυτών που δεν έχουν ψηφιακές ικανότητες. Ε, σημαντικό αυτό. Τώρα, τι, κάνουν, ε, τι κάνει η Άιζα σε σχέση με τις ανάγκες των κρατών μελών και κάποια παραδείγματα. Μπορούμε να αναφέρουμε π.χ. το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας ε, που είχε καθοριστεί ως ανακοίνωση της Κομισιόν. Δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα για την εφαρμογή του. 24 κράτη-μέλη το ε, μετέφεραν προσαρμόζοντάς το βεβαίως στις δικές τους ανάγκες γιατί το κάθε κράτος μέλος είναι διαφορετικό, είναι σαφές αλλά υπάρχει ένα κοινό όραμα μεταξύ αυτών των 24 μελών μια κοινή προσέγγιση. Αυτό λοιπόν είναι ένα καλό παράδειγμα μιας δράσης ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μας επιτρέψει να εργαστούμε με τον ίδιο τρόπο και την ίδια προσέγγιση. Κάτι το οποίο δεν σημαίνει πως βεβαίως ε, θα είναι τα πάντα όλο ίδια. Τώρα νομοθετικά κενά και τεχνικά ρυθμιστικά ζητήματα. Υπάρχει κάτι το οποίο προβλέπεται ήδη και συζητιέται και στο πλαίσιο του πακέτου της ε, ψηφιακής αγοράς που είναι η ε, επικαιροποίηση αυτής της στρατηγικής και του πλαισίου διαλειτουργικότητας για να λάβει υπόψη τα μαθήματα και τις ορθές πρακτικές των κρατών Και εδώ μπορούμε να προσθέσουμε την πρόταση του ΆΙΖΑ στο τετράγωνο που αφορά μια καινούργια αρχιτεκτονική. Οπότε έχουμε ένα πλήρες πακέτο στρατηγική, πλαίσιο, αρχιτεκτονική και χαρτογραφία. Μέρος ε, της πρότασης που έχετε μπροστά σας. προστασία των δεδομένων τώρα αναφέρεται ρητός στην πρόταση πως το πρόγραμμα ISA 2 πρέπει να ε, λάβει υπόψη τις ε, αρχές ε, της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων. Αυτό υπάρχει ως αρχή στην τρέχουσα πρόταση του του λεχθέντος πρέπει να αναφέρουμε, όπως είπα, πως εμείς δίνουμε κάποια συστατικά στοιχεία, προδιαγραφές, ορολογία που χρησιμοποιούνται για να δώσουμε λύσεις. Και σε τελική ανάλυση η ευθύνη βεβαίω ε, είναι των επιχειρήσεων που πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες και να εγγυηθούν όσοι ακολουθούν αυτούς τους κανόνες. Ναι, τα συστατικά στοιχεία πρέπει να λάβουν υπόψη, οπωσδήποτε, τη σχετική νομοθεσία, αλλά μετά αυτοί που θα τα χρησιμοποιήσουν πρέπει και αυτοί να λάβουν υπόψη τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι εταιρείε τώρα που προτείνουν δράσεις. Μία διευκρίνηση οι δράσεις που προτείνονται στο πρόγραμμα ΆΙΖΑ και ΆΙΖΑ 2 προτείνονται από διοικήσεις των κρατών μελών και τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Οπότε δεν λαμβάνουμε προτάσεις από τις εταιρείες. Η διαδικασία λοιπόν είναι πως επαφίεται στις διοικήσεις των κρατών μελών να προτείνουν κάτι. Οι δράσεις αυτές δεν σχετίζονται οπωσδήποτε με τις περιφέρειες. Δεν υπάρχει λοιπόν άμεση χρηματοδότηση των περιφερειών, δήμων, οτιδήποτε, αλλά τα αποτελέσματα μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν από εθνικές διοικήσεις και τα λοιπά. Μια τελευταία παρατήρηση. Οτιδήποτε γίνεται από το πρόγραμμα είναι στην διάθεση όλων των κρατών μελών και σε μια κοινή πλατφόρμα. Ήδη η πλατφόρμα περιέχει τα αποτελέσματα του προγράμματος ΆΙΖΑ όσον αφορά τις προδιαγραφές αλλά και τις λύσεις εκείνες οι οποίες ε, ε, έχουν ε, επιτευχθεί με τη στήριξη του προγράμματος αυτού. Και να τονίσω εδώ πέρα μια συγκεκριμένη περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που έχει υποστηρίξει το πρόγραμμα ΆΙΖΑ και έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από όλες τις ε, πρωτοβουλίες που έχουν υποβληθεί από τους οργανωτές. Όλες λοιπόν οι πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει χρησιμοποιούν αυτά τα οποία είχε ε, προτείνει το πρόγραμμα Άιζα. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την κυρία Ραβέλα Πεντρόζο από την Πορτογαλία. Ε, έχετε παρουσιάσει μία μελέτη για την Πορτογαλία. Έχετε λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ. Άκουσα όλους με προσοχή. Εγώ τρία μόνο ζητήματα θέλω να σας αναφέρω. Ανησυχίες ή, εν πάση ε, για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Η αίσθηση που είχα εγώ από το πρόγραμμα ΙΖΑ είναι ακριβώς αυτό που είπατε ορισμένοι, ότι δηλαδή εξαιρετικά τεχνικό, εξαιρετικά ε, ότι δηλαδή πολλά κρατημέλη συμμετέχουν αποκλειστικά για τα ίδια, ότι δηλαδή κινούνται, ότι είναι ένας άβλος κύκλος στην ουσία. Ε, πώς θα ανοίξει λοιπόν προς τους πολίτες και προς τις επιχειρήσεις. Τα τεχνικά ζητήματα, τα πρότυπα, τα PTI, η προστασία κτλ. αλλά Αυτά μπορούν να είναι ένα μπλοκ που μας ε, ε, απορροφά, αλλά κάποιες φορές ξεχνάμε γιατί υπάρχουμε. Και αν δεν θέλουμε να έχουμε το AZA 3, είναι απαραίτητο να φτιάξουμε μια νέα νοοτροπία που εξετάζει τι έχουμε κάνει, τι θα έπρεπε να κάνουμε και να δημιουργήσουμε αυτού του είδους ε, τις στιγμές για τα εθνικά κράτη-μέλη. Δηλαδή, Κάποιε φορέ το ερώτημα είναι ποιο είναι ο ρόλο τη Κομισιόν και ποιο είναι ο ρόλο του κράτου μέλου. Και όταν προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την μεταγραφή, συνήθω το κάνουμε με ρυθμιστικό τρόπο, αλλά δεν το κάνουμε με την οτροπία μας. Οπότε κάποιες φορές πρέπει, ε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα Γιατί πραγματικά δηλαδή φαίνεται να μην καταλαβαίνουμε, να μην συναισθανόμαστε ακριβώ ότι κάνουμε. Όμω, υπάρχουν αρκετά χρήματα και ο κόσμο δεν βλέπει κάποιο κομμάτι που να έχει ολοκληρωθεί και να αποδίδει. Το τρίτο στοιχείο που θέλω να τονίσω και που είναι κάτι που και στο παρελθόν συζήτησα πολύ με τη Μαργαρίδα γιατί γνωριζόμαστε εδώ και κάποια χρόνια. Πάντοτε το ζήτημα είναι το ίδιο. Δηλαδή όταν ε, βρισκόμαστε σε συνεδριάσεις ε, και είμαστε μαζί με τους εκπροσώπους των κρατών μελών κάποιες φορές ε, η ασκείται πίεση ε, στην ίδια αίθουσα. Δηλαδή, όταν όλα τα κρατήματα έχουν συμφωνήσει ότι το θέμα της διαλειτουργικότητας θα πρέπει να ε, απασχολεί μόνο τις κυβερνήσεις, κατάλαβαν ότι αυτό που κάνουν είναι το σωστό και ότι η κοινωνία δεν έχει καμία σχέση. Είναι κάτι που εμείς ένα μικρό κλαμπ κρατών μελών, μια λέσχη θα το χρησιμοποιήσει, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια γιατί εμεί είμαστε εκπρόσωποι του, των, των πολιτών, των λαών. Είναι κάτι το οποίο λοιπόν θα πρέπει να ε, σημάνει τη διαφορά για μας και για την Κομισιόν όταν μιλάμε για το ΙΖΑ 2 είναι το θέμα των τεχνικών ε, οικοδομικών λύθων. Ναι, είναι απαραίτητη. Αλλά η ένταξη όλων είναι ένα θέμα το οποίο δεν... ένταξη δηλαδή των πολιτών είναι κάτι το οποίο δεν συζητάμε αρκετά κατά τη γνώμη μου. Σας ευχαριστώ. Γκμόφσκι από, από την Πολωνία. Είστε τυχεροί λοιπόν που έχετε διαχειριστεί την ψηφιοποίηση. The Dziękuję ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως η συζήτηση που κάνω αυτή τη στιγμή ακολουθεί ενδιαφέρουσα κατεύθυνση, αλλά δείχνει και την πολλαπλότητα των ερωτήσεων και των ζητημάτων που αποδεικνύει σε ποιο βαθμό είναι περίπλοκος ο ψηφιακός κόσμος. Ορισμένοι είπαν Ε, και δεν έχουμε τονίσει αρκετά τον κίνδυνο του αποκλεισμού. Νομίζω πως όλο αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Είναι πολύ σημαντικό και φυσικά όποτε ε, ε, εντυπωσιαζόμαστε τόσο πολύ από νέες υπηρεσίες ή νέα επιτεύγματα, δεν καταφέρνουμε να καταλάβουμε ότι ε, δεν μπορεί όλος ο κόσμος να εκμεταλλευτεί και να υποφεληθεί από τις ψηφιακές υπηρεσίες. Και ελπίζω πως εδώ η τεχνολογία, είμαι βέβαιος πως η τεχνολογία θα μας βοηθήσει, διότι τα συστήματα γίνονται όλο ένα και πιο περίπλοκα και πιο εξελιγμένα, πιο προηγμένα. Ε, έχουμε δυνατότητες αναγνώρισης του εισφωνής. Ε, Είναι σημαντικό λοιπόν να ε, καταλαβαίνουμε και να σκεφτόμαστε τις δυνατότητες να οργανώσουμε μαθήματα, να, διδάξουμε τον κόσμο πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τις ψηφιακές υπηρεσίες ή διαφορετικά μπορούμε να αφήσουμε ταυτόχρονα ανοιχτούς τους ε, χάρτινους δρόμους, να μην ε, να, να, να λειτουργούν παράλληλα δηλαδή οι αναλογικές με τις ψηφιακές ε, λύσεις για κάποιο διάστημα. Το θέμα είναι ποιε λύσει θα χρησιμοποιηθούν περισσότερο και πού. Η ψηφιοποίηση έχει νόημα και η διαλειτουργικότητα έχει νόημα εφόσον έχουμε όλοι τα ίδια πρότυπα. Ε, και η διαδικασία θα πρέπει να είναι η εξή. Όταν λείπει η, η δυνατότητα ε, ή το πρότυπο να προσπαθούμε να βρούμε ε, κάποιο πρότυπο γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαφορετικά αν δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος μπορούμε να αφήσουμε περισσότερη ελευθερία ώστε όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται να μπορούν να επιλέξουν τις κατάλληλες λύσεις από μόνοι τους. Σε κάποιες από τις ομιλίες σας αναφέρετε την προστασία των δεδομένων που είναι νομίζω πολύ σημαντικό ε, θέμα Ξέρω πως πολλές άλλες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές το συζητούν, αλλά όταν μιλάμε για, την ε, για συμβιβαστικές λύσεις υπάρχουν και για ψηφιακή ε, αγορά υπάρχουν ένα σωρό παράμετροι. Κάτι ακόμα που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη είναι η κυβερνοασφάλεια. Νομίζω ότι στον κόσμο όπου ζούμε δεν υπάρχει τρόπος να αφήσουμε κατά μέρος την ε, ασφάλεια. Ε, θα πρέπει τα συστήματα να είναι ανοιχτά, ανοιχτά και προσβάσιμα στους πολίτες. Αυτό σημαίνει πως είναι προσβάσιμα και για τους, ε, για τους hackers, αυτούς που επιτίθενται στα δίκτυα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ σοβαρά και τις πτυχές ασφάλειας για να μπορούμε να την εγγυηθούμε. Ευχαριστώ. Και τώρα το επιστέγασμα της σημερινής απόψινής ακρόσης θα είναι ο κ. Ζωχίνιο. Πέντε λεφτά έχετε κ. Ζωχίνιο. Η απόψινή μας ε, συνεδρίαση δείχνει πως ε, οι τρόποι εργασία μας συγκλίνουν ώστε να βρούμε μία ή την καλύτερη δυνατή λύση. Οι εισηγητές μας ε, ήδη μας παρουσίασαν ένα πρώτο σχέδιο. Έχουμε και τροπολογίες, έχουμε συμφωνία με ε, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα έχουμε ένα μήνα για να παρουσιάσουμε και να ορίσουμε <laughs> και να συμπεριλάβουμε νέες τροπολογίες. Εγώ ορισμένα θα αναλάβω την πρωτοβουλία να τις συντάξω με βάση τα όσα μπόρεσα να αποκομίσω από την απόψινή συζήτηση. Επίσης γνωρίζουμε πως υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στην Ήτρε και ένα άλλο στην ΙΜΚΟ που είναι ε, συγχρονισμένα και ότι η ΛΥΜΠΕ θα, ε, θα αποβάλει τροπολογίες που θα εγγυάται ακριβώς, θα καλύπτει ακριβώς τις, ε, τα θέματα της ε, κυβερνοασφάλειας, της προστασίας των δεδομένων, χωρίς να ξεχνάμε αυτό που είπε η συνάδελφο Δάλη, ότι δηλαδή καλύτερο τρόπο για να τα επιτύχουμε την προστασία είναι να εγκρίνουμε το πακέτο για την προστασία των δεδομένων, που είναι ακόμα υπό εξέλιξη αυτή, αυτό το φάκελο. Τώρα, τα όσα μας εκθέσατε ε, και τα όσα μας αναπτύξατε απαντούν σε πολλά από τα ερωτήματα Ανάπτυξη λοιπόν μία κοινωνία ε, για όλους. Έχουμε τι τροπολογίε 1 μέχρι 15 σχεδόν ακριβώς στοχεύουν σε αυτό το θέμα της ε, καθολικότητας της καταπολέμησης ε, του ψηφιακού χάσματος, μείωση των δεφικών φραγμών. Επίσης εδώ ε, εννοείται και κάτι άλλο, αλλά καλύτερα είναι να το λέμε και πιο ξεκάθαρα στην τροπολογία 8, την ανησυχία δηλαδή της ανάπτυξης μιας κοινή σημειολογίας που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντική. Η Μαργαρίδα είπε ότι εμείς δίνουμε ε, τα θεμέλια, είπε foundations στα αγγλικά, αλλά ε, δίνουμε και τα τούβλα. Εγώ πιστεύω ότι ναι, πρέπει να φτιάξουμε τα θεμέλια. Είναι και ορισμένα επίσης βλάκια. Όχι όλα. Mm. Ε, κάτι θα τα πω μόνο πορτογαλικά γιατί αλλιώς δυσκολεύω τους διερμηνείς. Αλλά πάντως πιστεύω πω εδώ θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε το, να θέσουμε ένα όριο, δηλαδή ποιε είναι οι εφαρμογέ, ποιε είναι οι εφαρμογέ, οι εθνικέ και ποιε είναι για το ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιε μπορούμε να αφήσουμε στην κοινωνία ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί. Συμφωνώ να έχουμε τι ίδιε του κανόνε, να έχουμε προδιαγραφέ ασφάλεια κτλ. και κυρίως να εγγυηθούμε την διαλειτουργικότητα που είναι το θέμα κλειδί ολόκληρη αυτής της διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά, αυτό που ανέφερε η δόκτωρο Μαργαρίδα, που ήδη υπάρχει σε κάποια μορφή, είναι να ξέρουμε πόσες φορές έγινε όντως αυτό που μπορούσε να κάνει εκείνη. Πόσες φορές δηλαδή και πόσες διαδικασίες εξελίχθηκαν με βάση τα όσα υπάρχουν στην, πλατφόρμα και πόσες φορές αυτά αναπτύχθηκαν και αυτό πρέπει να το τονίσουμε ακόμη περισσότερο στην έκθεση Υπάρχουν ήδη δύο σχετικές ε, τροπολογίες, οι 17 και 25 που αναφέρονται σε αυτό το θέμα, καθώς επίσης και υπάρχει και κάτι ακόμα ε, το οποίο αναφέρθηκε και ανεπίσημα ότι όντως ε, η νέα θηρίδα για τις καλές πρακτικές θα πρέπει να είναι και πιο δραστήρια. Δηλαδή δεν, πρέπει, δεν αρκεί να ξέρουμε ότι υπάρχει, αλλά είναι καλύτερο να προχωρήσουμε και να κάνουμε μεγαλύτερη διάδοση των καλών πρακτικών. Και αυτό είναι σημαντικό και περιλαμβάνεται στις τροπολογίες 12 και 19. Στη συνέχεια έχουμε κάποιες τροπολογίες που έχουν σχέση με τη διαδικασία και αυτό ήδη ανεφέρθη από την Κομισιόν, δηλαδή διαδικασίες απλές που θα εγγυώνται όμως αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος Μαραγκάλ, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που να είναι μετρήσιμα Έχουμε 21, 22, 27 και 28 τροπολογίες που εν, απλοποιούν τις διαδικασίες, δηλαδή πότε χρησιμοποιούνται ε, οι πράξεις κατεξιοδότηση, η διαδικασία επίγουση κτλ. Τέλο πάντων διαδικαστικά ζητήματα. Στη συνέχεια είναι καλό να παροτρύνουμε τη συνεργασία ε, και κυρίως τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη και τους διοικητικούς μηχανισμούς της, της επιχειρήσης. Αυτά περιλαμβάνονται στην 13 και στην 23. Τώρα, αν από τώρα εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα όπως είπαμε και στην αρχική εισήγηση και θα ολοκληρώσω ήδη ξεπέρασα ναι. κατά 38 δευτερόλεπτα το χρόνο ομιλίες μου αλλά ε, να έχουμε δηλαδή δημόσιες υπηρεσίες, ε, εταιρείε και πολίτες, αλλά να έχουμε και, τα, να έχουμε και παράγοντες αξιολόγηση. Εδώ έχουμε την 11, 24 και 29 και τέλος μια, ένας προβληματισμός που είναι από τη ΛΥΜΠΕ και έχει να κάνει με την διαφάνεια και με την ασφάλεια της ενημέρωσης, που είναι η τροπολογία 18. Ε, είμαστε στην αρχή όμως της δουλειάς αυτής, έχουμε πολύ ακόμα δουλειά μπροστά μας που πρέπει να γίνει σωστά γιατί είναι σημαντική. Και αυτό χρειάζεται να ε, συνειδητοποιήσουμε ότι είναι σημαντική αυτή η δουλειά, ότι δουλεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση αλλά και θα πρέπει διαρκώς να τη βελτιώνουμε την εργασία μας. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι εσείς ξεκινήσατε με αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Είναι το 17ο προ σημείο της ημερησία μας διάταξης για σήμερα και θα ήταν φυσιολογικό ο κ. Μπόνι να ακολουθήσει μετά τη δική σας συμβολή ως σκιώδης εισηγητής από το ΕΛΚΑ. Κύριε Μπόνι, έχετε το λόγο. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλες οι τροπολογίες που πρότεινε ο Κάρλος είναι πάρα πολύ χρήσιμες και όλοι θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Βέβαια έχουμε ένα μήνα ακόμα στη διάθεσή μας για να κάνουμε και κάποιες επιπλέον. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στα εξή τέσσερα σημεία. Πρώτον, όταν μιλούμε για διαλειτουργικότητα, νομίζω θα είχε νόημα να διασυνδέσουμε πιο στενά τις προσπάθειες που καταβάλει το ευρωπαϊκό επίπεδο, που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο, με τις υφιστάμενες προτεραιότητες στα διάφορα κράτη-μέλη. Και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχει και ένα δεσμευτικό χαρακτήρα λίγο αυτό το ίσα 2, ότι ε, καλή συνεργασία, αλλά καλύτερη συμφωνία επί κάποιων προτεραιοτήτων. Δεύτερο σημαντικό για μένα. Πώς ελέγχεις ότι η αρχιτεκτονική και το πλαίσιο που προτείνεται σε αυτό το κείμενο για τη διαλειτουργικότητα θα είναι συμβατή με νέες προκλήσεις και με νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Τι εννοώ. Ας φανταστούμε μία κατάσταση που έχουμε ε, ηλεκτρονική υγεία στην Ευρώπη αυτό θα είναι ένα μοντέλο που θα επιτρέπει τη διασύνδεση σε όλα τα κρατη και είναι αρκετό και μπορεί να δεχθεί τις νέες λύσεις και τα νέα συστήματα. Γιατί τώρα είμαστε στο 2015 και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το 20. Μέχρι τότε ε, θα έχουν γίνει πάρα πολλά. Ε, είναι και πολλές οι νέες ε, τεχνολογίες και οι δέσμοι μέτρων για την ενιαία ψηφιακή αγορά που ε, εκπονεί αυτό τον καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να εγκρίνουν όλοι οι ενεχόμενοι. Όταν κληθούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα θα δούμε ότι υπάρχουν και νέες δυνατότητες και νέες προκλήσεις. Άρα και εδώ θα πρέπει να χωρούν αυτές και να υπάρξει ε, πρόβλεψη για αρκετή ε, διαλειτουργικότητα που να είναι συμβατή με τις νέες αλλαγές στην τεχνολογία. Το επόμενο τρίτο θέμα έχει να κάνει με το εξής. διάφορες απειλές και πώς μπορούμε να αποφύγουμε επικαλύψεις και ε, δίπλο δουλειέ ουσιαστικά ανάμεσα στο πρόγραμμα αυτό και όσα κάνουν τα κράτη-μέλη από την πλευρά τους που δραστηριοποιούνται και αυτά στο κλάδο. Θα δω πώς θα συντάξω τις τροπολογίες μου σχετικά. Πιθανότατα να χρειαστεί και πάλι δέσμευση και υποχρεωτική συμμετοχή όλων των ενεχομένων στην ετήσια αναθεώρηση. Ξέρω ότι αυτό είναι λίγο διοικητικό κορσές και βάρος, αλλά αν θέλουμε να αποφύγουμε τις επιπλοκές, μάλλον πρέπει να βρεθεί μια λύση, να τη βρείτε. Και ένα τελευταίο, τέταρτο, βεβαίως αυτό δεν έχει να κάνει ακριβώς και άμεσα με το έγγραφο που συζητούμε εδώ και τώρα, αλλά αυτό το περίφημο νομοθετικό χάσμα που αναφέραμε. Νομίζω θα πρέπει να έχουμε και τα δύο ταυτόχρονα ή σε αντίστοιχο χρόνο ας πούμε. Ε, να το εγκρίνει αυτό το κοινοβούλιο και να έχουμε και καλή γνώση για το τι συμβαίνει στην κάθε νομοθεσία και τι αλλαγές χρειάζονται. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει. από τη διευκρίνηση του νομικού πλαισίου και της νομικής βάσης στην οποία βρισκόμαστε. Είναι συμπληρωματικό και μόνο αυτό και ευχαριστούμε Κάρλος για το πνεύμα σου και την ενέργεια που αφιερώνεις σε αυτή την υπόθεση γιατί μας κάνεις όλους να καταλαβαίνουμε καλύτερα και με νέο βλέμμα και μια φρέσκα και ματιά έχει καταφέρει να μετατοπιστεί η συζήτηση από την αυστηρά τεχνική στην ουσιαστική και στον πυρήνα πραγματικά που πρέπει να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόιρε έχει αποχωρήσει. Ο κύριος ε, Μαραγάλα, λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τώρα ορισμένα πράγματα να επιμείνουμε σε κάποιες έννοιες. Σας είπα εμείς πώς θα προχωρήσουμε τη μέθοδο. Είναι καταπληκτική και πολύ συναρπαστική αυτή η προσπάθεια. θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή επικουρικότητα απέναντι στην συγκέντρωση θα πρέπει ε, να το συγκεκριμενοποιήσουμε αυτό γιατί τα κριτήρια και οι κανόνες είναι πολύ γενικοί και μάλιστα εκ των προτέρων έτσι, να φροντίσουμε να συνοδεύουμε, να βοηθάμε τα κράτη-μέλη ε, που κάνουν τα πρώτα τους βήματα τώρα στη διαλειτουργικότητα αυτή. Στη συνέχεια. Το θέμα αυτό της διαφάνειας του ανοιχτού χαρακτήρα, της διάβγειας για τις λύσεις που προτείνονται θα πρέπει επίσης να κυριαρχεί και να βελτιώσουμε τα αποτελέσματά μας. Να είμαστε κατακαιρματισμένοι ή ανταγωνιστικοί στην αποτελεσματικότητα. Γιατί αυτό θα είναι η εις της διαλειτουργικότητας. Από εκεί θα κριθεί η επιτυχία του προγράμματός μας. Και η απόδειξη θα είναι ότι δεν θα χρειαστεί ένα ίσα τρία, όπως είπα προηγουμένως. Το θέμα του συντονισμού τώρα και της συλλογική δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Στα πλαίσια του ψηφιακού θεματολογίου δεν θα ήταν, πιστεύω, ε, παραδεκτό να έχουμε μόνο μια κάθετη ανάλυση της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης για το ΙΣΑ αλλά θα πρέπει να εντάσσεται ε, σε μια εγκάρσια προσέγγιση ε, για να αξιοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις λύσεις που έχουμε την οικονομία κλίμακας με άλλες οργανικές δομές και υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με συνεργασία και συλλογική, αποτελεσματική όμως και ουσιαστική δράση. Ε, θα ήταν πάρα πολύ καλό αυτό εντάξει, έχουμε το χρόνο να κάνουμε τροπολογίες, προτάσεις και ε, με θετικό πνεύμα να προχωρήσουμε και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά τη συμφωνία με την γραμματεία θα διαβάσω τα όσα ε, λέει εδώ πέρα η κυρία Ματίας. Το πρόγραμμα ΆΙΖΑ, διαλειτουργικές λύσεις για τις ευρωπαϊκές ε, δημόσιες διοικήσεις, πλησιάζει το τέλος του. 31 Δεκεμβρίου 2015, οπότε απαιτείται ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αφορά την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών δημοσίων διοικήσεων και εστιάζει σε θέματα όπως η διαλειτουργικότητα, η διασυνοριακή, η διαλειτουργικότητα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προμήθειες, τιμολόγια, ανοιχτά δεδομένα, το δίκτυο, συμμετοχικά εργαλεία και πλατφόρμες με στόχο τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ως ε, υπερασπιστές της διαφάνειας και ποιοτικής λειτουργίας του δημοσίου τομέα και συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων ψηφιακών υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν ειδικά τους πολίτες που ζουν μακριά από τα κέντρα των πόλεων σε γενικές γραμμές είμαστε υπέρ του προγράμματος αυτού για έναν εξεχρονισμό που θα βασίζεται στην πληροφορική. Τώρα ήρθε η ώρα της Κομισιόν. Η κυρία Ίγκεστατ, ίσως εκπρόσωπος ε, της Γενικής Διεύθυνσης Digit. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, να πω πως αναφερθήκατε στον ρόλο της ε, Κομισιόν εδώ πέρα και ιδιαίτερα στην αρχή της επικουρικότητας ε, και στην συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Κομισιόν Φτερού. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ξανά πως ε, λαμβάνουμε κάποια μέτρα για να είμαστε συντονισμένοι στο πως ε, συνεργαζόμαστε σε διαφορετικά προγράμματα και έχουμε δέσμευση από όλες τις ε, υπηρεσίες για αυτό το θέμα και όπως είπε και η κυρία Γεωργίευα Προσφάτως στην Υπουργική Διάσκεψη στη Ρώμη στις 3 Δεκεμβρίου η Κομισιόν είναι έτοιμη να βοηθήσει να στηρίξει στον επιθυμητό βαθμό, στο βαθμό που επιθυμούν τα κρατημέλη, στον εξυγχρονισμό των δημοσίων διοικήσεων. Συγκεκριμένα για το ΆΙΖΑ έχουμε την ίδια πρόθεση, συνεργαζόμαστε με τα κρατη για να ε, επιτύχει το πρόγραμμα ΆΙΖΑ. Αλλά βεβαίω ε, είναι πολύ σημαντική και η ρόλη του καθενός. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στην Μαργαρίτα για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, που ακούστηκαν. Ναι, ίσως αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Μαργάλ να αναφέρω κάποια ζητήματα που είναι ανοιχτά. Πρώτα απ' όλα η φήμη της Κομισιόν για το πρόγραμμα ΆΙΖΑ. Ο αρμόδιος είναι ο Επίτροπος Έτιγκερ και ο Αντιπρόεδρος Έντσιπ. Όπως ήδη νομίζω αναφέρθηκε. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα του πώς τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν καλύτερα την δουλειά τους. Ε, τώρα δεν είναι δουλειά της Κομισιόν να παρέμβει, αλλά το γεγονός πως υπάρχει καλύτερη ευελιξία και συντονισμός μεταξύ των διαφόρων πολιτικών οπωσδήποτε θα είναι κάτι το θετικό για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στον συντονισμό τους. Η άλλη ερώτηση που αναφέρθηκε αφορούσε ακριβώς την ανάλυση της ε, χρηματοδότησης. Υπάρχει ε, μπορούμε να σας απαντήσουμε και λεπτό Όσον αφορά τώρα τα μαθήματα κλειδιά. Όλα αυτά τα οποία μάθαμε και βρίσκονται στην πρόταση αυτή βασίστηκαν στις προτάσεις που υπάρχουν στην ενδιάμεση αξιολόγηση, στην έκθεση εφαρμογής και στις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη της διοικής των, των κρατών μελών, της Κομισιόν. Όσον αφορά τώρα τα κενά στην νομοθεσία. Ε, είναι κάπως πιο δύσκολη αυτή η ερώτηση. Ήδη έχουμε μια πιο σαφή άποψη των νομοθετικών κενών. Τώρα δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορούμε νομίζω να δούμε, γιατί το ζήτημα αναφέρθηκε και από την Επιτροπή Άιζα το τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή αυτή τη ε, στιγμή. Θα το δούμε μαζί τους. Οπωσδήποτε η αναθεώρηση του πλαισίου της στρατηγικής και της αρχιτεκτονικής, αλλά τώρα αν υπάρχουν κενά δεν μπορώ να πω σε αυτή την φάση. Είναι κάτι που θα συζητήσουμε οπωσδήποτε με την Επιτροπή και ελπίζω να επανέλθουμε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Τώρα ήρθε η ώρα του εισηγητή. Κύριε Τωρίνιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε πάλι το λόγο. Δεν χρειάζεται να κάνω κατάχρηση. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είμαστε σε ένα σημείο όπου μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε συζητήσει για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με τους διάφορους σκιώδεις. Το μόνο που μπορώ να προσθέσω τώρα είναι να βεβαιώσω ότι είμαστε σε σωστή, στην κατάλληλη φάση για να ξεκινήσουμε το δρόμο και θέλω και πάλι να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Ευρωκοινοβούλιο καταρχήν διότι ε, διοργάνωσε αυτή την ακρόαση και δεύτερον όλους όσους ε, την μετέτρεψαν σε τόσο πολύ ενδιαφέρουσα ε, ακρόαση του εμπειρογνώμονε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέλη τη ΣΥΤΡΙ και του συναδέλφου συνεισηγητέ και όσου ήταν παρόντε απόψε. Έχουμε λοιπόν τα κατάλληλα στοιχεία για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. Ευχαριστώ. Και τώρα βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση, όλους όσοι μίλησαν σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και ε, πληροφοριών. Ιδιαίτερα δε θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας με πρώτο τον εισηγητή τον κύριο Ε, Φυγητή για αυτό το σημαντικό θέμα και την τόσο ε, κρίσιμη έκθεση. Πρέπει να σας πω τώρα ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λίγη στις 26 Φεβρουαρίου του 2015 για το σχέδιο γνωμοδότησης. To, uh, go forward. Έχουμε ένα μήνα καιρό και φαντάζομαι ότι θα αποκρισταλωθούν στις τροπολογίες τα όσα εδώ συζητήσαμε. Και ένα τελευταίο που έχω να σας πω είναι η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης 26 Φεβρουαρίου 2015 στις 3 ώρα στις Βρυξέλλες. Είναι έκτακτη αυτή η συνεδρίαση. 26 Ιανουαρίου, συγγνώμη, 23 Φεβρουαρίου στις 3 και πάλι στις Βρυξέλλες κανονική συνεδρίαση. Δύο ημέρες, 23 και 24 Φεβρουαρίου. Στις 24 είναι στις 9 η ώρα το πρωί. Αυτές είναι οι προσεχείς μας συνεδριάσεις. Στην ίδια αίθουσα πιθανότατα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Καλό σας βράδυ και καλή σας όρεξη.